Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι η ψηφοφορία θα γίνει μετά από τα δύο θέματα συζήτησης που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Την επιστολή του Αλεξάνδερ Λάμστορ που ήταν επικεφαλής της Αποστολής Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη 25 με 27 Μαρτίου φέτος και θα ήθελα να του δώσω το λόγο να μας παρουσιάσει τα απορίσματα της αποστολής. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πληροφορήσω τους συναδέλφους για την επίσκεψη που έκανα ως επικεφαλής της ομάδος αξιολόγησης των εκλογών. Οι εκλογές θα γίνουν τον Ιούλιο. Κύριε, είναι κάπως παράξενο να πάει κανείς τον επόμενο χρόνο τον Μάρτιο. Έγινα τον Ιούλιο, συγγνώμη. Αλλά ουσιαστικά ήταν μια ε, επίσκεψη μετά από την παρουσίαση της τελικής έκθεσης που έκανα τον Νοέμβριο και μετά έγινε η επίσκεψή μου για να δω τι συνέχεια δόθηκε στα διάφορα θέματα. Νομίζω ότι λειτουργήσαν όλα πολύ καλά σε γενικές γραμμές. Η κατάσταση στη Λιβύη είναι ακόμα πολύ ασταθής. Έχουμε έλλειψη πλήρους ε, ασφάλειας εκτός σε κεντρικό επίπεδο και οι πολιτοφυλακές εξασκούν την εξουσία ουσιαστικά σε περιφερειακό επίπεδο και δεν ξέρει κανείς πώς θα εξελιχθούν τα θέματα αυτά στον τομέα της ασφαλείας και αυτό είναι ένα τμήμα της αλήθειας και της πραγματικότητας. Η, δεύτερη όμως πτυχή είναι ότι δεν υπήρξε κάποια σοβαρή αντίδραση σε πολιτικό επίπεδο, Η σε επίπεδο ασφαλείας. Η διαδικασία μετάβαση είναι βραδύ, αλλά πηγαίνει προ τη σωστή κατεύθυνση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα όταν αντιμετωπίζουμε τι εξελίξει στη Λιβύη. Γιατί μετά από εννέα πια μήνες έχουν γίνει πολύ λίγα πράγματα σε ό,τι αφορά τη συνταγματική διαδικασία, παραδείγματο χάρη, που ήταν το κύριο θέμα για μένα στη δική μου ημερήσια διάταξη όταν ήμουν εκεί. Σίγουρα έχει εξανεμιστεί ο ενθουσιασμό ο οποίο είχε διαφανεί στι εκλογέ πέρσι τον Ιούλιο. Δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλέ στο Κοινοβούλιο. Αυτό δεν είναι βέβαια απαραίτητο για μια χώρα σε μετάβαση, αλλά υπάρχει γενική εντύπωση ότι το Εθνικό Συνέδριο θα πρέπει να προχωρήσει περισσότερο τα πράγματα. Και η διαδικασία του συντάγματος μπορεί να φαίνεται απόμακρη από την καθημερινή ζωή, αλλά παρόλα αυτά δημιουργεί μεγάλο ενδιαφέρον μεταξύ των πολιτών. Είναι κάτι για το οποίο θέλουμε να επιτευχθεί πρόοδος και αν θυμόσαστε ότι η χώρα είναι διηρημένη σε τρεις περιφέρειες που στέλνουν 20 άτομα η κάθε περιοχή σε μια συντακτική συνέλευση και αυτό έχει αποφασιστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά δυστυχώς αναρωτιόμαστε γιατί δεν έχει γίνει κάτι για αυτά τα πράγματα, γιατί ο κύριος στόχος αυτού του Εθνικού Συνεδρίου να δημιουργήσει την επιτροπή η οποία θα εκπονήσει το Σύνταγμα. Και υπάρχει μια ασάφεια για τη σύνθεση αυτής της επιτροπής. Δεν θα σας πω τις λεπτομέρειες, αλλά μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει κάτι τέτοιο, όταν έχουμε μια κατάσταση όπου ο λαός περιμένει ότι θα ψηφίσει στις εθνικές εκλογές για να υπάρξει σύνθεση της συντακτικής συνέλευσης και από την άλλη πλευρά υπάρχει μια νομική αντιμετώπιση που προβλέπει την, το διορισμό αυτής της Επιτροπής που θα εκπονήσει το Σύνταγμα από το τωρινό Κοινοβούλιο. Το ε, Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την προηγούμενη απόφαση και μπορεί τελικά το Εθνικό Συμβούλιο να ακολουθήσει την οδό του διορισμού. Ίσως με τον τρόπο αυτό σε επίπεδο ικανότητος, με το διορισμό να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την ικανότητα αυτών των ατόμων, αλλά βέβαια μόνο με τις εκλογές μπορούν να έχουν την απαραίτητη δημοκρατική νομιμοποίηση. Η μετάβασή μου στη Λιβύη <clears throat> ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Ήταν να υπάρχει μια κόπωση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρα πολλέ αντιπροσωπείε τη Ευρωπαϊκή Ένωση πήγαν εκεί, μείνανε για δύο-τρει μέρε. Χρησιμοποιούν του πόρου τη αντιπροσωπεία και των κρατών μελών. Αλλά τουλάχιστον οι ΜΚΟ με τι οποίε συνεργαζόμαστε μα υποστήριξαν ιδιαίτερα και είχαμε πολύ καλέ συναντήσει μαζί του και ιδίως γιατί ενδιαφέρονται και εστιάζουν περισσότερο στο πώς να προχωρήσει η πολιτική διαδικασία στη Λιβύη. Και πέραν τη κόπωση που ανέφερα προηγουμένω σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι υπάρχουν σαφεί ευκαιρίε για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να συνεχίσει την συμμετοχή τη στη διαδικασία αυτή. Αυτό το οποίο κάναμε ήταν να προσπαθήσουμε να φέρουμε μαζί όλου του εμπλεκομένου στην συνταγματική αυτή διαδικασία και μα είπαν όλοι αυτοί που προσκαλέσαμε και ήρθαν και είχαμε καλή προσέλευση ότι ήταν η πρώτη φορά που όλοι αυτοί είχαν βρεθεί στην ίδια αίθουσα. Ήταν κάτι το οποίο με εξέπληξε ιδιαίτερα, γιατί τα Ηνωμένα Έθνη έχουν μια πολύ μεγάλη ε, αντιπροσωπεία στη Λιβύη, κάνουν πολύ καλή δουλειά σε πάρα πολλά θέματα, αλλά για τη συνταγματική διαδικασία θα πρέπει να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αυτή η οποία έδωσε την ουσιαστική όθηση. Και ήταν από τις συναντήσεις που είχαμε ότι όλε αυτέ οι συναντήσει θα μπορούσαν να ήταν πολύ πιο μακροσκελεί από ό,τι προβλεπόταν, γιατί ήταν τόσα πολλά τα θέματα που είχαμε να συζητήσουμε. Αυτό το οποίο τώρα προέκυψε από τι συζητήσει είναι ότι υπάρχει ευρεία συνένεση ότι το μελλοντικό σύνταγμα θα πρέπει να βασίζεται στον Ισλαμικό νόμο, στη Σαρία, σε οποιαδήποτε από τι πολλέ ερμηνείε τη. Δεν κοιτάζουμε μονάχα το τμήμα του ποινικού δικαίου που έλκεται από τη Σαρία. Αλλά η χώρα αυτή βλέπει τον εαυτό της ως μια Ισλαμική χώρα η οποία πρέπει να αντιμετωπίσει με αυτόν τον τρόπο τον εαυτό της. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε πώς αυτό μπορεί να είναι συμβατό με τα δικαιώματα των μειονοτήτων, τα ατομικά δικαιώματα και όλα αυτά. Αυτό είναι κάτι το δεν έχει συζητηθεί αυτή τη στιγμή, γιατί η συνταγματική διαδικασία είναι μόνο στο σημείο της εκκίνησής της. Δεν είναι ακόμα σαφές με ποιο τρόπο η χώρα αυτή θα μπορέσει να ενσωματώσει τις υποχρεώσεις της βάσης του διεθνούς δικαίου στο εθνικό της, στην εθνική της συνταγματική διαδικασία αν η πηγή του συντάγματος είναι η Σαρία, τότε ο εθνικός νόμος είναι μια πηγή δικαίου, αλλά και οι διεθνείς συμβάσεις θα πρέπει να είναι μια πηγή δικαίου. <clears throat> Έχουμε συζητήσει και για το Ιράκ σαν ένα υπόδειγμα σε σχέση με τα θέματα αυτά. Η, η Αίγυπτος δεν ήταν τόσο ενθαρρυντική σε σχέση τη συνταγματική διαδικασία. Αυτά τα οποία γίνονται λοιπόν στη Λιβύη ξεκινούν τώρα μόνο και γι' αυτό είναι πολύ θετικό που μπορέσαμε να είμαστε παρόντες και που μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Όχι φυσικά για να ηγηθούμε τη συζήτηση, αλλά για να πληροφορήσουμε καλύτερα με τις ε, γνώσεις και την εμπειρία που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τέτοιες μεταβατικές διαδικασίες. Τέλος πρέπει να πω ότι η χώρα αυτή έχει ευτυχώς μια εκλογική επιτροπή η οποία έχει πετύχει πολύ ψηλό επίπεδο απόδοσης ήταν πάρα πολύ και εκπληκτικά ουσιαστικά ικανοί και καλά οργανωμένοι αυτοί που διοργάνωσαν τις εκλογές τον Ιούλιο πέρσι. Υπάρχει αυτή η Επιτροπή βέβαια, δεν έχει ακόμα επίσημο χαρακτήρα, αλλά όσο δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει μια εκλογή για τη συντακτική συνέλευση, είμαστε στο κενό. Γιατί χρειάζεται ένας εκλογικός νόμος εάν γίνει με ψηφοφορία η επιλογή της συντακτικής συνέλευσης. Χρειαζόμαστε ένα μήνα για να γίνει κάτι τέτοιο. Ενώ λοιπόν η πρόοδος είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, τα πράγματα πηγαίνουν αργά. Αλλά σας λέω και πάλι πολύ καλή εκλογική επιτροπή. Εν κατακλείδη. Θα πρέπει να παραμείνουμε παρόντες και να συμμετέχουμε στη διαδικασία, αλλά με ένα τέτοιο τρόπο, ο οποίος βοηθάει τους Λίβιους για αυτό το οποίο χρειάζεται. Όχι να πηγαίνουμε και να ξαναγυρίζουμε στην Ευρώπη και να μην δίνουμε συνέχεια. Χρειαζόμαστε οργανώσει οι οποίε θα είναι έτοιμε να έχουν μια συνεχή παρουσία. Ευτυχώ υπάρχει ένα ευρύ φάσμα διεθνών φορέων ΜΚΟ με τι οποίε συνεργαζόμαστε. Υπάρχουν πολύ ισχυρέ τοπικέ ε, ΜΚΟ που συμμετέχουν πλήρω σε αυτέ τι διαδικασίε. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να συμμετέχουμε και να είμαστε παρόντες και έχουμε και την έκθεση της Επιτροπής αξιολόγηση των Εκλογών που περιέχει σημαντικές και ενδιαφέρουσες συστάσεις και έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία που μπορούμε να δώσουμε στους Λίβιους. Κλείνοντας, η κατάσταση της ε, αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάπως ε, δύσκολη κατάσταση, έφυγε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ο οποίο να εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ πιστεύω πρέπει να υπάρξει μια στεναρή παρουσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με το αντίστοιχο επίπεδο υψηλών επιπέδων προσωπικού είναι μια χώρα που βρίσκεται στη γειτονιά μας. Ξέρω ότι όταν ο, ήταν ο Καντάφης στην εξουσία δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής η Τριπολίτιδα, αλλά είναι μια χώρα εν μεταβάση που θα είναι πάρα πολύ σημαντική για μας για πολλά θέματα και γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε να τι υποστηρίζουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής διαδικασίας με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως θα πρέπει να καλύψουμε την ηγεσία της αντιπροσωπείας. Αν υπάρχουν ερωτήματα, είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, είσαστε πραγματικά σαφέστατο και καλύψατε όλα τα θέματα. Δεν έχει ζητήσει κανεί το λόγο για ερωτήσει. Τουλάχιστον δεν είδα να ζητάει κανείς το λόγο. Και άρα θεωρώ ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό και να περάσουμε πάρα αυτό στο επόμενο θέμα, όπου και πάλι έχω την χαρά να σου δώσω το λέγω, γιατί πρόκειται για τη σύσταση προ το Συμβούλιο σχετικά με την 68η Σύνοδο τη Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ. ή στο εισηγητή. Έχετε λοιπόν και πάλι το λόγο. Ähm, Πολύ ωραία. <laughs> Να μιλήσω γερμανικά. Γιατί ο πρόεδρος μας δεν έχει πρόβλημα με τα γερμανικά. στην ομάδα εργασίας για τα Ηνωμένα Έθνη σε ό,τι αφορά τη σύσταση προς το Συμβούλιο. Πρόκειται για ένα καλό κύκλο εργασιών. Δίνουμε εγκαίρως την κοινοβουλευτική μας ε, άποψη. Στις 7 Μαρτίου έγινε εκτεταμένη συζήτηση με τον επικεφαλής πολυμερών σχέσεων και ε, διακυβέρνησης, Κριστίνε Περόν. Ήταν λοιπόν πάρα πολύ παραγωγική αυτή η συζήτηση, αυτή η συνεδρίαση. Η σύσταση κυκλοφόρησε στην ομάδα εργασίας. Σήμερα θα παρουσιαστεί εδώ στην Επιτροπή και θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Τις τροπολογίες ε, θα πρέπει να τις ε, έχουμε λάβει μέχρι τις 18 Απριλίου από σήμερα. Φέτος δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εσωτερικό του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και στα θέματα ειρήνης και ασφάλειας αφενός, αλλά και αφετέρου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Rule of law. Ένα βασικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση έχει έξι τμήματα, δεν πρόκειται να σας τα παρουσιάσω όλα. Για να μην ε, επιβαρύνω τους ε, συναδέλφους. Είναι αρκετά συνοπτική η έκθεση, μπορείτε να τη διαβάσετε. Το πρώτο θέμα που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιο φορέα. Καλεί τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τις αντιπροσωπείες να φροντίσουν ότι υπάρχει πραγματικά ε, συνεκτικότητα και έμφαση σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη. Να τονίσουμε ποια ήταν, η πρόοδος που πετύχαμε και πού θέλουμε να συνεχιστεί η πρόοδος. Θίγουμε και θέματα μεταρρύθμισης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ένα θέμα το οποίο τα τελευταία χρόνια θεωρείται ότι δεν έχει κινηθεί προς τα εμπρός, αλλά αντιθέτως έχει κάνει βήματα προς τα πίσω. Και γενικώ υπάρχει μια, μια αντιστατικότητα να συζητιέται το θέμα αυτό. Και αυτό αφορά ε, κάποιες χώρες που θέλουν να έχουν μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας, όπω η Βραζιλία για παράδειγμα, αλλά και άλλε χώρε. Το θέμα αυτό λοιπόν το συζητήσαμε. Θα σα ενημερώσουμε. Η μακροπρόθεσμη, ο μακροπρόθεσμο στόχο μια Ευρωπαϊκή έδρα εξακολουθεί να αποτελεί θέση και του Κοινοβουλίου αλλά και διαφόρων κρατών μελών. Αλλά φυσικά δεν έχουμε, δεν τρέφουμε αυταπάτες. Ένα δεύτερο κρίσιμο ζήτημα είναι το θέμα της ε, ευθύνη για προστασία, responsibility to protect. Θα πρέπει να, να μην παρανοείται η έννοια αυτή. Πρόκειται για ένα... Δεν πρόκειται για στρατιωτική παρέμβαση, μιλάμε για πρόληψη, για προστασία της κοινωνίας των πολιτών, την πρόληψη ε, εμπόλεμων ε, συγκρούσεων, πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια για αυτούς που θέλουν. Αυτός ο ευρύτερος ορισμός λοιπόν της ευθύνης για προστασία είναι κάτι το οποίο υπογραμμίζουμε και αναφέρουμε δύο χώρες, την Συρία και το Μάλι, δεν σας προκαλεί έκπληξη. Δύο χώρες για τις οποίες ε, τοποθετήθηκε με έντονο τρόπο ο Γενικός Γραμματέας. Σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουμε κυρίως ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πρόθεσή του σε όλους τους τομείς της εργασίας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και σε ό,τι αφορά την ε, ενίσχυση της καθολικής διαδικασίας ε, αναθεώρησης και κυρίως ε, τονίζουμε την πρόσβαση των μη κυβερνητικών οργανώσεων στις διαδικασίες αυτές σε ό,τι αφορά και για παράδειγμα την ελευθερία έκφρασης και εδώ αναφέρω για παράδειγμα τη συμμετοχή των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα. Έχουμε επίσης αναφέρει θέματα για το κρατός δικαίου. Όπως σας είπα, υπήρξε μια, το Σεπτέμβριο του 2012 μια συζήτηση υψηλού επίπεδου για το θέμα αυτό και απευθύνουμε σύσταση προς το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Ένα θέμα το οποίο πάντα προκαλεί δυσκολία στη Νέα Υόρκη πώς εργάζονται και συνεργάζονται οι κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια σε ό,τι αφορά παγκόσμια θέματα. Δηλαδή, η εκτελεστική εξουσία έχει δικαίωμα δράσης, ε, αλλά το κοινοβούλιο είναι αυτό το οποίο νομιμοποιεί την εκτελεστική εξουσία και μπορεί να συνδράμει στην εκτελεστική εξουσία. Αλλά στη Νέα Υόρκη είναι πάντα δύσκολο να συζητιούνται τέτοια θέματα ε, και είχε προβλεφθεί κάτι τέτοιο για την 68η Σύνοδο, αλλά τελικά δεν πρόκειται να συζητηθούν αυτά τα θέματα αυτά. Οι συνάδελφοι εδώ στο Κοινοβούλιο τάσσονται υπέρ μια κοινοβουλευτική συνέλευση ε, των Ηνωμένων Εθνών και άλλοι, όπως εγώ, θεωρούν ότι δεν θα, υπήρξε, δεν θα υπήρχε οποιαδήποτε προστιθέμενη αξία σε μια τέτοια κοινοβουλευτική συνέλευση. Θα ήταν στην καλύτερη περίπτωση μια συνέλευση πάρα πολλών ε, ατόμων που δεν θα είχαν όμως οποιαδήποτε νομιμότητα. Δεν πρόκειται να εκδημοκρατιστεί τίποτα. Αλλά παρόλα αυτά γίνεται και πάλι όπως κάθε χρόνο μια τέτοια συζήτηση γιατί πολλοί συνάδελφοι έχουν αντίθετη άποψη και χαίρομαι και προσβλέπω στις μελλοντικέ συζητήσεις προβλέπεται ψηφοφορία στις 30 Μαου προκειμένου τον Ιούνιο να περάσει το θέμα αυτό στην Ολομέλεια για να ψηφιστεί. Ευχαριστούμε πολύ, λέγει ο Πρόεδρος. Και τώρα να δώσω το λόγο στο σκιώδη ηγητή από το ΕΛΚ, τον κύριο Πρέντα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας τον συνάδελφό μας, Γκρανφ Λάμστορφ, για την ε, ποιότητα του εγγράφου που εξεπώνησε. Εκφράζω και τη λύπη μου, διότι δεν μπορούμε να εγκρίνουμε το έγγραφό μας ε, γρηγορότερα. Πολύ πιο πριν την διεξαγωγή της 68ης Γενικής Συνελεύσεως. Έχω κάποιες ιδέες για το έγγραφο. Θα τις διαβιβάσω μέσω τροπολογιών. για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου. Συμφωνώ να τα αναφέρουμε αυτά, αλλά θα πρέπει να αναφερθούμε και στη δημοκρατία και όπου αναφέρονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, στο κείμενο εγώ θα υποβάλω τροπολογία για την προσθήκη και της λέξεως δημοκρατία σε αυτά τα σημεία. Συλλογική προσπάθεια θα πρέπει να καταβληθεί στο 1C, αλλά σε κάποιες περιστάσεις θα πρέπει κανείς να δραστηριοποιείται χωρίς ε, συνένεση. Και το Μάλι ήταν ε, μια τέτοια περίσταση που το δείχνει, δείχνει αυτή την ανάγκη. Στο 1Ι, στο σημείο αυτό, δεν συμφωνούν τα κράτη-μέλη. Δεν συμφωνούν όσον αφορά την έδρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Θα πρέπει όμως να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να δουν το ζήτημα μακροπρόθεσμα. να κινηθούν προς την ιδέα μιας έδρας ενιαίας Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για το 1F, ενίσχυση του ρόλου και του κύρους της Γενικής Συνελεύσεως των Ηνωμένων Εθνών και στο L για την Συρία ε, θα πρέπει να αναφέρονται τα ανθρωπιστικά δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα όλοι οι εμπλεκόμενοι στο, στην κρίση θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο 1M που αφορά το Μάλι νομίζω ότι πέρα από τις στατιωτικές πτυχές της κρίσης θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και τη δημοκρατική μετάβαση και την πολιτική διαδικασία. Σχετικά με το εμπόριο όπλων, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τη συμφωνία που επετεύχθη την περασμένη εβδομάδα. Που είναι αποτέλεσμα ετών διαπραγματεύσεων. Στο σημείο π ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα έπρεπε να είναι ένας μοχλός για την περιοδική αναθεώρηση σε σφαιρικό επίπεδο και εν τέλει το Συμβούλιο θα πρέπει να μας ενημερώσει, να υποβάλει μια έκθεση για την Γενική Συνέλευση. Όλες αυτές τις ιδέες θα τις συμπεριλάβω ε, σε διάφορες τοπολογίες θα υποβάλω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρέντα. Τελευταία παρέμβαση η κυρία Μουνίθ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να συγχαρώ τον κύριο Λάμστορφ όχι μονάχα για την έκθεσή του αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο διεύθυνε την ομάδα εργασίας και τον τρόπο με τον οποίο είχε επαφές με τους εκπροσώπους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα Ηνωμένα Έθνη και με όλη την ομάδα που ασχολείται για τα θέματα των Ηνωμένων Εθνών. Ε, επανέρχομαι σε αυτά που είπε ο κύριο Πρέντα προηγουμένως για την ανάγκη το Συμβούλιο να πληροφορήσει το Κοινοβούλιο για τη συνέχεια που δίδει στις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αλλιώς, καταλήγουμε σε μια κατάσταση όπου εμείς εκδίδουμε κάθε χρόνο διαφορετικές συστάσει και σε πολλές περιπτώσεις δεν προκύπτει απολύτως τίποτα. Αναγκασόμαστε να επαναλαμβάνουμε τα ίδια στοιχεία και πολλές φορές έχουμε και διαφορετικές διεκδικήσεις που αλλάζουν συνέχεια τα πράγματα. Χρειάζεται να έχουμε μια μεγαλύτερη συνέχεια σε σχέση με τις διεκδικήσεις και αυτά που ζητάμε από τα κράτη-μέλη στα Ηνωμένα Έθνη ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προς την κατεύθυνση αυτή Θέλω να σταθώ μονάχα σε ορισμένα σημεία, τα οποία θα οδηγήσουν σε τροπολογίε. Καταρχήν το θέμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση σαν παίκτη στο συνολικό, στο παγκόσμιο στερέωμα. Εκεί δεν είχαμε πολλά αποτελέσματα. Είναι απαραίτητο να υπάρχει μια μεγαλύτερη συνέχεια στην εκπροσώπηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στι ομάδε G στο σύστημα των, και στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών στην Γενική Συνέλευση, στην 67η και 7 Γενική Συνέλευση, Υπήρχε προηγουμένως μία αμνία για αυτή την παρουσίαση, για αυτή την παρουσία και τη συνέχεια που, να έχει, που έχει εξαφανιστεί από το εφετινό έγγραφο χωρίς να έχουμε πετύχει κάποια αποτελέσματα στο παρελθόν. Για το Συμβούλιο Ασφαλείας ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η θέση των κρατών μελών, αλλά ξέρουμε και ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενεκρίθη κατ' επανάληψη για την έκθεση για την πολυμερή αντιμετώπιση στο διεθνή χώρο και αναφέρεται ο στόχο να υπάρξει μια έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα μακροχρόνιο στόχο, μακρόπνο στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό ανεξάρτητα από τη θέση των κρατών μελών που φυσικά δεν συμφωνούν όλα με μια τέτοια ρύθμιση. Στα θέματα ασφαλείας θα πρέπει να επανέλθουμε στο ψήφισμα 325 του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ε, διάσταση του φύλου σε σχέση με την πρόληψη συγκρούσεων και την ανθρωπιστική βοήθεια καθώς και τις ενέργειες αφοπλισμού και ε, επανενσωμάτωσης των πολιτοφυλακών στην κοινωνία. Και επίσης για το εμπόριο όπλων, και εδώ θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια επικαιροποίηση με την συμφωνία που επετεύχθη στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Επίσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, νομίζω ότι θα πρέπει να επαναλάβουμε και πάλι <clears throat> μια αμνία στην ε, απόφαση των ΗΠΑ το 2005 για τα θέματα διαφθοράς, όπου θεωρήθηκε ότι η διαφθορά είναι μία μορφή παραβιάσεως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γι' αυτό θα πρέπει να ζητήσουμε από, τον, ε, από την, από την ύπατη εκπρόσωπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο να θεσπίσει ένα σχέδιο δράση για να εφαρμοστούν τα συμπεράσματα της Σύμβασης των για τη διαφθορά και επίσης να παρακολουθηθεί η κατάσταση της εφαρμογής αυτής της σύμβασης σε επίπεδο μονογραφής, υπογραφής, επικύρωσης στα κράτη-μέλη <clears throat> και να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα αυτά στα Ηνωμένα Έθνη. Υπάρχουν ορισμένες τροπολογίες που θα παρουσιαστούν από την πολιτική μου ομάδα, από τον Γιώ Λάινεν και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικές και τις υποστηρίζω πλήρως. Το να θεωρηθούν τα εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας το να υπάρξει ένα πλαίσιο για, τον κολλασμό αυτών των εγκλημάτων κατά του περιβάλλοντος όπως και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, η ενίσχυση της ικανότητας εργασίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και εν γέννη η ενίσχυση σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον για πιο με πιο συγκεκριμένο τρόπο από ό,τι περιλαμβανόταν στην αρχική έκθεση πάση περιπτώσει θα τα καταθέσουμε όλα αυτά με τη μορφή τροπολογιών και καλή επιτυχία στον κύριο Λάνστορ. Σας ευχαριστώ. Αλεξάνδρε, θες να πεις κάτι σχετικά? Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, για τα ευγενικά λόγια που είπαν οι συνάδελφοι για το έργο μου και φυσικά είναι απόλυτα ορθό να κατατεθούν και τροπολογίες μετά από αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Είπε ο Κριστιαν Πρέντα ότι είναι σημαντικό το θέμα της δημοκρατίας και φυσικά ισχύει αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια εμεί έχουμε προσπαθήσει να εστιάσουμε στο θέμα αυτό της υποστήριξης της δημοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο και επομένω θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα θέματα του κράτους δικαίου έχουν μια μεγάλη προβολή. Ε, και νομίζω ότι το κράτος δικαίου θα πρέπει να παραμείνει η κύρια εστίαση για τα θέματα αυτά. Για το Μαλή φυσικά πρέπει να υποστηρίξουμε τη δημοκρατική μετάβαση. Αυτά που είπε ο Κρίστιαν και η Μαρία επίσης είναι ότι φυσικά πρέπει να υπάρξει αυτή η επικαιροποίηση με την τελευταία απόφαση των Ηνωμένων Εθνών για το θέμα της εμπορίας όπλων. Εδώ δεν υπάρχει προφανώς καμία αντίρρηση. Θα γίνει αυτή η ενημέρωση του κειμένου για να λάβει υπόψη και αυτή την ε, απόφαση, κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό. Πιστεύω τώρα ότι η θέση των κρατών μελών μας για τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας συγκεκριμένα η Γαλλία αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο εμείς ως ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν την αποδεχόμαστε γιατί εμεί θέλουμε μια έδρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό θα πρέπει να οδηγήσει και σε μια γενικότερη μεταρρύθμιση της σύνθεσης του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δεν μπορεί να είναι μια μεμονωμένη αλλαγή, αλλά θα πρέπει να συνδεθεί με ε, άλλες αλλαγές και όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν σε ένα ορίζοντα ενό ή δύο ετών αλλά σε ένα ορίζοντα 5-10 ετών όπου εμεί θα πρέπει να επανεξετάσουμε το σύνολο των θεμάτων που έχουν να κάνουν με την ε, σύνθεση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Για τι τροπολογίε του Γιολάιν, αν κατάλαβα καλά, πρόκειται για το να θεωρηθούν τα εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος ότι είναι εξίσου σοβαρά και εξίσου κολάσιμα με τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε και εγώ χαίρομαι για την ευκαιρία να επανέλθουμε στο θέμα αυτό στην επόμενη συνάντησή μας, στην επόμενη συζήτησή μας για τα θέματα αυτά. Υπάρχουν κάποια δικήματα κάτω του περιβάλλοντος τα οποία μπορούν να έχουν αυτό το χαρακτήρα κατά την άποψή μου. Επομένως, προσβλέπω στην ε, περαιτέρω συζήτηση, χαίρομαι για τις τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τα διεκπαιρεώσουμε όλα αυτά τα θέματα για το χρονοδιάγραμμα, όπως είπε και ο κύριος ε, Πρέντα. Εγώ περιμένω από τη γραμματεία να μας πει πότε προβλέπετε να έρθουμε στην Ολομέλεια. Εγώ θα ήθελα το ταχύτερο να το να διεκπαιρεώσουμε αυτά τα θέματα, αλλά νομίζω ότι η γραμματεία μπορεί να κάνει καλύτερα διαχείριση των θεμάτων αυτών. Ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρε. Να σας πω τώρα. Προθεσμία είναι 18 Απριλίου, 5η στις 12 οι και όχι 11. Θυμηθείτε όχι 11 Απριλίου. 18 Απριλίου. Άννα, θες να πάρεις το λόγο για αυτό το θέμα. Ορίστε. Απλώς να υποστηρίξω ένθερμα αυτά που είπε ο Αλεξάνδρ Λάμστορφ για το ρόλο του Κοινοβουλίου που πρέπει να απευθύνει έκκληση και να θέτει στη συζήτηση το θέμα μιας έδρασης Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτό είναι κάτι πραγματικά σημαντικό. Να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι στο παγκόσμιο προσκήνιο φορέας αν δεν ζητήσει μεταρρύθμιση του Συμβουλίου και συνεπώς να αποκτήσει δική της έδρα Ευρωπαϊκή Ένωση στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Και έχει τεράστιες δυνατότητες αυτό να οδηγήσει σε μια μεταρρύθμιση που ιδαλλιώς ποτέ δεν θα γινόταν. Και να υποστηρίξω αυτό που έλεγε η Μαρία Μουνίθ για την ανάγκη να αναφερθούμε στην σύμβαση του ΙΕ κατά της διαφθοράς και την ανάγκη τα κράτη-μέλη μας να εφαρμόσουν αυτές τις διατάξεις και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Μία από τις συστάσεις της συμβάσεως του ΙΕ κατά της διαφθοράς αφορά την ποινικοποίηση του παράνομου πλούτου. Είναι ένας τομέας που ήταν πάρα πολύ δύσκολος και στις χώρες μας και παρά το γεγονός που όλοι παρακολουθούμε το πώς η χρηματοστική και οικονομική κρίση σχετίζεται άμεσα με τα επίπεδα της διαφθοράς που έχει διαδοθεί ε, ανάμεσα στους πολιτικούς που επηρεάζονται από τα οικονομικά συμφέροντα, γι' αυτό υπάρχει και αντίθεση στην ποινικοποίηση του παράνομου πλουτισμού. Αυτό ταιριάζει με αυτά που συνεπέρανε η Επιτροπή μας ΚΡΙΜ και με αυτά που η Επιτροπή Ντρουά συνεπέρανε. Άρα δεν θα πρέπει να διστάσουμε, θα πρέπει συγκεκριμένα, σαφώς να το διατυπώσουμε αυτό και να το υποβάλουμε στην προσοχή του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Γκόμες. Εδώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και μπορούμε να πάμε στη ψηφοφορία για το σχέδιο ψηφίσματος για την έκθεση προόδου για το 2012 για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η συγκητής είναι ο κ. Ρίτσαρτ Χάουιτ. Κύριε Χάουιτ, θέλετε να πείτε κάτι πριν την ψηφοφορία. Να είμαι πάρα πολύ σύντομο. Ε, να πω τρία πράγματα. Καταρχάς, ε, θα θυμάστε, φίλοι, Θα θυμάστε ότι αναβάλαμε σκόπιμα την ψηφοφορία λόγω της πολιτικής κρίσης ε, στα Σκόπια. Και ο κύριος ε, Μπούζεκ που είναι εδώ πέρα και χαιρόμαστε που είναι εδώ πέρα ως πρώην ε, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμετείχαμε σε μια αποστολή που ενθαρρύναμε τις πολιτικές διαπραγματεύσεις στα Σκόπια και θα γνωρίζετε πιο πολύ εξ ότι ήταν ε, επιτυχής η αποστολή αυτή και υπήρξε συμφωνία μεταξύ ε, των ε, μερών, των πολιτικών δυνάμεων της χώρας χωρίς μετά από ολοκλήρωση της έρευνας των περιστατικών της 24 Δεκεμβρίου στη χώρα και να πω και προς τον Πρόεδρο και στον Πρόεδρο Μπρόκ ότι ήταν σωστή απόφαση της Επιτροπής να αναβληθεί η ψηφοφορία και νομίζω ότι αυτό ενθάρρυνε το σωστό και θετικό αποτέλεσμα. Απέστειλα το κείμενο στα μέλη της Επιτροπής. Προγραμματιζόταν λοιπόν να γίνει η ψηφοφορία σήμερα και να γίνει η ψηφοφορία σε ένα επικοδομητικό πλαίσιο. Πλαίσιο τονίζω. Και είμαι βέβαιος ότι τα μέλη ε, σκοπεύουν να τηρήσουν τη συμφωνία αυτή. Να τονίσω επίσης ότι ο δεύτερος ε, γύρος των εκλογών έλαβε χώρα χτες στη χώρα αυτή και υπάρχουν κάποια αποκρατατικά αποτελέσματα τα οποία και διάβασα με προσοχή και είμαι βέβαιος ότι και άλλοι θα το έκαναν αυτό πριν ε, από τη σημερινή ψηφοφορία. Και τέλος να σας υπενθυμίσω ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος στο πλαίσιο ε, της διαπραγματεύσεων την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσει την ε, ενδιάμεση αναθεώρηση, τη σχετική έκθεση για την ενδιάμεση αναθεώρηση στο Συμβούλιο, άρα θεωρώ ότι είναι πολύ έγκαιρη η χρονική συγκυρία ε, για την ψηφοφορία. Σε ό,τι αφορά τους εμβιβασμούς, ε, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε λεπτομερή ανάλυση τους κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, αλλά να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που καταλήξαμε σε μια ναι. σχετικά γρήγορη συμφωνία για πολιτικά πολύ ευαίσθητα ζητήματα. Να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές ομάδες και πιστεύουμε ότι έχουμε ε, καλά προγνωστικά και νομίζω ότι στο σημείο αυτό μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, να σας συγχαρώ να συγχαρώ και τον πρόεδρο Μπούζεκ για την επιτυχία τους ε, μαζί με τον ε, Επιτροπό σε ό,τι αφορά την επίσκεψή σας στα Σκόπια και σε ό,τι αφορά την άρση των φραγμών, των πολιτικών φραγμών μεταξύ των δυνάμεων των πολιτικών στη χώρα. Πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία... Να δώσω το λόγο στην κυρία Γιαννάκου. Κύριε Πρόεδρε, να αποσύρω την τροπολογία με υπαριθμό 44. Θέλω. Αποσύρω την τροπολογία 44. Okay, it's noted. Μάλιστα το σημειώσαμε. Στην τρίτη σελίδα. Δεύτερη σελίδα, τρίτη σελίδα, λέει ο πρόεδρο. Όχι. Ο κ. Κουματσάκο, έχει ζητήσει το λόγο. Πρόεδρε, ε, η, έκθεση, η ψήφιση για την έκθεση αναβλήθηκε λόγω των ε, ε, πολιτικών εξελίξεων στην ε, χώρα την οποία σήμερα εξετάζουμε στην έκθεσή μας και θα ψηφίσουμε. Ήθελα να ρωτήσω το Προεδρείο αν αυτή η πρακτική αποτελεί προηγούμενο και για άλλες εκθέσεις που θα, τυχαίνει να εξετάζονται ή να ψηφίζονται σε εποχή που χώρες οι οποίες θα αφορούν τις έκθεση βρίσκονται σε κάποια πολιτική αβεβαιότητα ή αν υπάρχουν αρνητικές εξελίξεις. Αποτελεί προηγούμενο, είναι μια ad hoc πρακτική. Και σε άλλες, το ξαναλέω, αν και σε άλλες εκθέσεις που αναφέρονται σε συγκεκριμένες χώρες, αν εκείνη τη στιγμή που έχει προγραμματιστεί ψηφοφορία, υπάρχουν εξελίξεις σε αυτές τις χώρες, αρνητικές, πολιτικές εξελίξεις, θα αναβάλλονται οι ψηφοφορίες μέχρι οι εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις να ομαλοποιούνται. Φτιάξαμε λοιπόν, μια προ... Ε, λοιπόν με αυτή την έκθεση ένα προηγούμενο. Φτιάξαμε ένα προηγούμενο, είναι ερώτηση προς το Προεδρείο. Κύριε Κουμουτσάκη, νομίζω ότι είμαστε πολιτικοί θεσμικοί, θεσμοί εδώ και αν έχουμε πολιτικά ζητήματα επί των οποίων έχουμε συμφωνήσει, μπορούμε να προχωρήσουμε βάσει των συμφωνιών μας. Θέλετε και εσείς το λόγο, κύριε Αλεξάνδρα ναι, ναι, ναι, δύο θέματα. Αφενό, νομίζω ότι δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο όταν οι πολιτικέ ομάδε συμφωνούν ότι η πολιτική κατάσταση σε οποιαδήποτε χώρα ε, καλό θα ήταν να αναβληθεί να γίνεται κάτι τέτοιο. Αυτό μπορεί να το αποφασίσει η Επιτροπή. Και το δεύτερο θέμα είναι μια ερώτηση προ τον Ρίτσαρτ ε, για την τροπολογία 1, όπου μιλάμε για την Μακεδονία ω το επίθετο και για το επίσημο όνομα. Γιατί, γιατί δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει πολιτικό υπόβαθρο, είναι θέμα διατύπωσης. Ο Πρόεδρος, κοιτάξτε τώρα, είμαστε στο θέμα της ψήφης. Έχουμε περάσει στην ψηφοφορία, στα αγγλικά. Ναι, λάβαμε πριν από μία ώρα εδώ τι τις προφορικές ε, τροπολογίες ε, και τις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες. Για πρώτη φορά λοιπόν βλέπω την τροπολογία υπαρθμών 1. Μπορεί να είναι εντάξει, αλλά γιατί. Γιατί είναι πολιτικό το θέμα είναι συντακτικό θέμα διατύπωσης. Οι συμβαστικές ε, τροπολογίες, λέει ο Πρόεδρος, είναι ε, μετά από συμφωνία των πολιτικών ομάδων. Να σας απαντήσει ο εισηγητής. Να είμαι σύντομος. Ο Αλεξάνδερ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι αυτό αποτυπώνει αυτά που συμφωνήθηκαν πέρσι. Ο κίνδυνος με το κείμενο αυτό είναι να φανεί ότι το Κοινοβούλιο τίθεται και υποστηρίζει μία πλευρά στο θέμα του ονόματας και κάποιοι θέλουν να χρησιμοποιηθεί όσο πιο πολύ γίνεται η ονομασία πρώην Γηκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και άλλοι θέλουν να χρησιμοποιηθεί ο όρος Μακεδονία Μακεδονικός. Άρα, εγώ πέρσι, προκειμένου να φτιάξω ένα κείμενο ισορροπημένο, τελικά καταλήγουμε να εκνευρίζουμε και τις δύο πλευρές. Και άρα, συμπεριλαμβάνουμε το επίσημο όνομα σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αλλά και μία φορά στο κείμενο χρησιμοποιούμε τον όρο Μακεδονικός, το οποίο μα το ζητεί, ζητά πολλοί κόσμος ε, από τη χώρα το οποίο αναφέρεται και σε ό,τι αφορά τη χώρα και σε ό,τι αφορά τη γλώσσα. Με την μία και μοναδική αυτή αναφορά ε, δεν αναζωπυρώνουμε την ε, διαμάχη. Το κάναμε και πέρσι, το κάνουμε και φέτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ και Χόιτ. Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να ξανακινήσουμε τη ψηφοφορία. την ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 Περνάμε τώρα στην τροπολογία 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Την 71. You're in favor against? Against. One more against. Close the vote. Yeah, it's adopted. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με 28 ψήφους υπέρ. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 75 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβιβαστική 8 με προφορική τροπολογία 2 και στην προφορική τροπολογία έχουμε μία προσθήκη η οποία έχει την έγκριση του εισηγητή. Να σας τη διαβάσω την πρόταση προφορικής τροπολογίας μετά την πρώτη ε, ε, πρόταση αναφέρεται ε, ότι προτείνει να υπάρχουν μελετές σχέσεις με τις όμορε ε, χώρες. Αυτό έχει συμφωνηθεί με τον εισηγητή. Να το ψηφίσουμε αυτό λοιπόν. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται με τις προφορικές τροπολογίες. Και τώρα περνάμε στην τροπολογία 76 υπέρ. Κατά, άποχες. Κατά παρακαλώ, δεν είδα. Κανείς κατά. Έγκρινεται λοιπόν. Η 9, συμβαστική 9, υπέρ. Συγγνώμη, συγγνώμη. Η 182, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 80, υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά την 80. one Εγκρίνεται. Συμβαστική εννέα, Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 88. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πάλι πρέπει να ελέγξουμε. 81 ηλεκτρονικά. Please close the vote. It's rejected. Απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ταυτόσιμες τροπολογίες 94, 95, 96 και 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 100 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της 100. Απορρίπτεται. 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 ο εισηγητής ο κ. Χάουιτ μια στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σε επαφή με τη Γραμματεία σήμερα το πρωί και πρότεινε μια τεχνικής φύσεως βελτίωση του κειμένου και την υποβάζω του προφορική τροπολογία και διαβάζω. Δεν πιστεύω ότι είναι πολιτικά επίμαχο θέμα. Αφορά τη σωστή απεικόνηση. νέα διατύπωση θα λέει. Καλωσορίζει τη συνεχής προσπάθειας για την πρόθεση νομοθετικού πλαισίου για, την πιλο... για τις διοικητικές διαδικασίες του πολιτικού ιδιωτικού τομέα, κυρίως όσον αφορά το νόμο για διοικητικούς υπαλλήλους και το νόμο για γενικές διοικητικές διαδικασίες. Και νομίζω ότι είναι σωστή η κατονομασία των νόμων και μετά συνεχίζουμε στο αρχικό κείμενο και λέμε καλή περαιτέρω προσπάθεια να γίνουν για να εγγυάται τη διαφάνεια, μεροληψία και επαγγελματισμό τη δημόσια διοίκηση, όταν να εξασφαλίζεται η πρόσληψη με βάση τα προσόντα και να ενισχυθεί είναι ήδη στο κείμενο. Αυτές οι πρώτες τρεις γραμμές να τις επαναλάβω, αυτές προτείνονται. Εντάξει. Όχι, όχι, είναι εντάξει. Δεν υπάρχει κανείς στις εναντίον της προφορικής τοπολογίας. Ψηφίζουμε 117 όπως είχε προταθεί, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 121 υπέρ κατά αποχές δεκτή 1.22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ κατά αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε εδώ ηλεκτρονικά. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Με μία ψηφοδιαφορά μονάχα. Συμβαστή 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστή 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Σύμβαστη 16 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 147 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 151 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, εγκρίνεται συγγνώμη 152, 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά μπορούμε να κάνουμε έλεγχο αν θέλετε. Πέρας. Ναι, ναι, απορρίπτεται. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 163 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 164 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 166 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε έλεγχο, 166. 166 ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. Για 166. 167. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 170 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 171 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 172 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 173 υπέρ. Κατά αποχές. Πάλι πρέπει να ελέγξουμε. 173 ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 174 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 175 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 199 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 5 υπέρ αποχές δεκτή. 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 9 <clears throat> υπέρ κατά αποχές δεκτή, Απολύτω, συγγνώμη, 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 13 υπέρ Όχι, δεν θέλουν οι σοσιαλιστές να ψηφίσουμε μαζί. 13. Υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 14 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 3 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται και αυτή. Τελική ψηφοφορία τώρα ηλεκτρονικά. Άρχεται ψηφοφορία. Ένα συνάδελφο ακόμα δεν έχει ψηφίσει. Γίνεται δεκτή με 38 ψήφους υπέρ, 39 υπέρ, 13 κατά και ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον εισηγητή τον κύριο Χάουιτ για την πολύ καλή εργασία σας. Πέρα ψηφοφορίας. είναι αυτό. Colleagues, let us start our uh, debate. Συνάδελφοι, ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με την παρουσία του κυρίου Ρωμάνο Πρόντι, ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΑ για το Σαχέλ. Θα συζητήσουμε για την κατάσταση στην περιοχή. Όπως ξέρετε, πέσει το Σεπτέμβριο ανακοίνωσε ο ΟΗΑ τη στρατηγική του για την ε, περιοχή του Σαχέλ. Γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δική τη στρατηγική για το Σαχέλ που χρονολογείται από το 2010 νομίζω. Αναπόφευκτο λοιπόν ότι πρέπει να εναρμονίσουμε τις δύο στρατηγικές. Έχω τη χαρά να σας ανακοινώσω ότι λόγω της πρωτοβουλίας του συναδέλφου του κυρίου Παντζέρη που είναι πρόεδρος της αντιπροσωπείας για την περιοχή μας συνοδεύουν εδώ οι πρόεδροι της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Αλγερίας, ο κ. Μπενκασέμ του Μαρόκου, ο κ. Κεμπερί και της Τινησίας ο κύριος Αμπτελραχήμ και ο κύριος Ακάμπη από τη Λιβύη έπρεπε να ακυρώσει την ε, έλευσή του την τελευταία στιγμή. Ακύρωσε την έλευσή του. Ο κύριος Μπροκ, ο πρόεδρος της Επιτροπής, έχει κολλήσει σε κυκλοφοριακή συμφόρηση κάπου στη Γερμανία λόγω της ε, λαμπρής οικονομικής αστιότητας της Γερμανία. Αν ήταν εδώ θα είχε αρκετό χρόνο να έρθει χαλαρά και ωραία λόγω της κρίσης. Εκτός όλων αυτών, θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Πρόντι να ξεκινήσει τη συζήτησή μας παρουσιάζοντας την κατάσταση για ένα δεκάλεπτο και μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση. Έχετε το λόγο κύριε Πρόντι. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ που με καλέσατε και με κάποια συγκίνηση επιστρέφω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με κάνει να ξαναζώ τα χρόνια της νεότητας σχεδόν. Απόψε έχω αυτά τα λίγα λεπτά για να σας παρουσιάσω συντομότατα την κατάσταση που επικρατεί στο Σαχέλ με ιδιαίτερη αναφορά ε, στο τι γίνεται τώρα, με ευρύτερο ε, απέρα από το Μαλί. Το Σαχέλ είναι τεράστια περιοχή, εκτείνεται από τον Ατλαντικό ωκεανό και φτάνει μέχρι την Ερυθρέα, συμπεριλαμβάνει πάνω από 5.000 χιλιόμετρα έχει πλάτος, ε, μήκος και 1.000 χιλιόμετρα πλάτος. Έχουμε τη Μαυριτανία, τον Μπουρκίνα Φάσο, τον Ήγυρα, το Τσάτ και το Μαλί. Αυτές οι πέντε χώρες συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη λωρίδα και το Μαλί είναι στο επίκεντρο της ε, προσοχής μας. Θα ήθελα καταρχάς να πω καταρχάς ότι πάντα ασχολούμουν με τα θέματα της ειρήνης. Πρέπει να πω ότι από την αρχή ήταν σαφές ότι η γαλλική παρέμβαση έγινε με τρόπο που ήταν εντελώς απαραίτητος διότι είχε σχεδόν καταρρεύσει η χώρα όταν οι ακρεφνείς ομάδες κινήθηκαν προς τον Νότο, προς τον Μπαμάκο, ήταν αναπόφευκτη αυτή η γαλλική παρέμβαση. Αυτό σίγουρα έλυσε ένα μέρος των προβλημάτων η γαλλική παρέμβαση, αλλά προφανώς δεν έχει επιλύσει την άλλη πτυχή της οργάνωσης μελλοντικής τη μη στρατιωτική πλευρά του ζητήματος του Σαχέλ. Η Γαλλία προβλέπει να αποσυρθεί και να αφήσει ευθύνη για τη σταθερότητα της χώρας σε κάποια δύναμη και συζητείται λοιπόν στο μέλλον πώς θα αντιμετωπιστεί το στρατιωτικό πρόβλημα στην περιοχή. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο στατιωτικό όπως προανέφερα, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστεί και η πολιτική πτυχή και ιδιαίτερα για τους πληθυσμούς του Βορρά, που επί μακρόν αισθάνθηκαν περιθωριοποιημένες και πολιτικά και οικονομικά. Και εμείς θα πρέπει συνεπώς από την αρχή να ξεκινήσουμε μια διαδικασία συμφιλίωσης που έγινε προσπάθεια πολλές φορές γι' αυτό κατά το παρελθόν. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα μόνο σημερινό, αλλά είναι ένα πρόβλημα που έχει ρίζες στο μακρινό παρελθόν. Και θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα διαπραγματευτικό τραπέζι το ταχύτερο δυνατόν, αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει να δώσουμε εγγυήσει ότι από τη στιγμή που οι διαπραγματεύσεις θα έχουν πετύχει αποτελέσματα, αυτά τα αποτελέσματα μετά θα εφαρμοστούν στο μέλλον. Και στις δύο προηγούμενες περιστάσεις υπήρξε συμφωνία, μετά όμως δεν υπήρξε καμία δυνατότητα ή βούληση να ε, δοθεί συνέχεια στις συμφωνίες, να εφαρμοστούν οι συμφωνίες. Ο οδικός χάρτης, το roadmap λοιπόν, για να φτάσουμε στη συμφωνία, έχει ξεκινήσει η κατάρτιση του οδικού χάρτη. Προβλέπονται νέες εκλογές τον Ιούλιο που μας έρχεται. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες για να συμβεί αυτό, αλλά πρέπει αμέσως να ξεκινήσει η διαδικασία για να είναι εφικτές οι εκλογές. Ο Ιούλιος είναι μια εποχή συχνά δραματική περίοδος διότι υπάρχουν μετεωρολογικά προβλήματα, η μετεωρολογική κατάσταση δυσκολεύει τις λύσεις. Αλλά η διεθνής κοινότητα θα πρέπει όμως να ξεκινήσει, να ξεκινήσει ε, αυτή την εκλογική διαδικασία, ούτως ώστε να διεξαχθούν το ταχύτερο δυνατόν ε, εκλογές. Σας έλεγα ότι αυτό εντάσσεται σε ένα πρόβλημα ανάπτυξης του Σαχέλ, που είναι ένα από τα πιο φτωχά μέρη του κόσμου αν πάρουμε την ταξινόμηση του κατακεφαλήν εισοδήματο των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο, βλέπουμε ότι οι χώρες του Σαχέλ είναι ανάμεσα στις τελευταίες χώρες σε αυτή την ταξινόμηση, με προβλήματα όπως είναι η ξηρασία και η έλλειψη τροφίμων. Εμείς στον ΟΗΕ έχουμε θεσπίσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική που εδράζεται τεσσάρων πυλώνων βασικών. Τον πρώτο τον ανέφερα για το πρόβλημα της ειρήνης και της ασφάλειας στο Μαλί. Δεύτερος πυλώνας είναι το πρόβλημα της σταθερότητας, της ανθρώπινης ούτως υπήν σταθερότητας, των ανθρωπιστικών προβλημάτων που δημιουργούνται και είναι η κληρονομιά αυτών των συγκρούσεων. Τεράστιο αριθμό προσφύγων που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι τεράστια η διάσταση του προβλήματος. Είναι 400 με 500 χιλιάδες τα άτομα τα εκτοπιστέντα, displaced, που έφυγαν από το σπίτι τους, είτε για να πάνε στο νότο του Μαλή, είτε να πάνε σε γειτονικές χώρες. Και τέλος, αυτό που απασχολεί περισσότερο τη στρατηγική μας είναι η μέσο μακροπρόθεσμη ανάπτυξη ε, αυτής της περιοχής. Μία ανάπτυξη που δεν μπορεί να περιορίζεται σε μεμονωμένες χώρες. Το πρώτο πρόβλημα είναι αυτό που είπε και ο γραμματέας του ΟΗΕ. Να καταλάβουμε ότι καμία χώρα από αυτές δεν μπορεί να αναπτυχθεί απομονωμένα. Και δεύτερον, Ποτέ δεν υπήρξε αναπτυξιακή στρατηγική συντονισμένη και συνδυασμένη ανάμεσα στις διάφορες χώρες αυτές. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται αναπτυξιακό σχέδιο συντονισμένο μεταξύ όλων και γι' αυτό ξεκινήσαμε μια δουλειά που δεν βασίζεται επί επιβολής εκ των άνω, αλλά έχουμε κινητοποιήσει τα πανεπιστήμια στην περιοχή. Ε, γίνονται οι πρώτες συνεδριάσεις και προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε την κατεύθυνση ανάπτυξης. Γεωργία, άρδευση, χρήση των υδάτων, συντονισμός των υποδομών, σχολεία, υγεία και ανάπτυξη της ενέργειας, ενεργειακών πηγών. Ε, αποκεντρωμένη ηλεκτροδότηση για τους πολίτες της περιοχής. Αυτό βέβαια απαιτεί συνεργασία όλων των δωρητών, των donors του κόσμου. Ξεκίνησα εγώ ε, προσκύνημα στις μεγάλες χώρες ε, για να συμβεί αυτό και στις δωρητές χώρες και βρήκα μεγάλη ευαισθητοποίηση λόγω του κοινού φόβου μάλιστα έναντι της τρομοκρατίας. Είναι η πρώτη φορά που η διεθνής κοινότητα Καταλαβαίνουμε τι έγινε στο παρελθόν. Ήταν, στο Ιράκ ήταν διερεμένη, στο Αφγανιστάν ήταν διχασμένη η παγκόσμια κοινότητα, στη Λιβύη ήταν διερεμένη, στη Συρία. Στο Σαχέλ όμως είδα ότι υπάρχει μια κοινή βούληση των κρατών για να μην εδραιωθεί σε αυτή την περιοχή η τρομοκρατία, μια βούληση δηλαδή, να γίνει κάτι. Η διεθνής κοινότητα προφανώς θα πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτή τη θετική τάση και θα ήθελα να κλείσω αυτή την σύντομη παρέμβασή μου όχι με μια στιγμή αισιοδοξία, αλλά λογική θετική τοποθέτηση. Δηλαδή η Αφρική δεν είναι πλέον η Αφρική του παρελθόντος. Βλέπουμε κάποια στοιχεία που δεν βλέπουμε κατά το παρελθόν. Το πρόβλημά μας στο αντικειμενικό δεν είναι να πετύχουμε αδύνατα, ανέφικτα αποτελέσματα, αλλά να φροντίσουμε ούτω ώστε το Σαχέλ να μπορεί να έρθει πιο κοντά μας. Να συνεργαστεί στα πλαίσια μιας απαρχής αφρικανικής οικονομικής ανάπτυξης. Είναι συγκεκριμένος ο στόχος, σαφής και ίσως μπορούμε να μπούμε και σε λεπτομέρειες αργότερα στο τι μπορεί να κάνει η διεθνή κοινότητα, τι διαθέτει η, Ευρωπαϊκή, η διεθνής κοινότητα για την ανάπτυξη. Ποια ήταν η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την οικονομική ανάπτυξη και που δεσμεύτηκε να δώσει και στο μέλλον. Μπορούμε να δούμε όλους τους ρόλους που μπορούν να παιχθούν στο παγκόσμιο προσκήνιο για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε Πορόντι μαζί με τον κύριο Ντανζό, ο οποίο είναι ο πρόεδρος τη Υποεπιτροπή για τα θέματα ασφάλειας. Γύρισαμε από το Μαλί και τον Ήγηρα το Σάββατο μόλι και μπορούμε να σα διαβεβαιώσουμε ότι η κατάσταση είναι πολύ πιο πολύπλοκη από ό,τι φαίνεται από την Ευρώπη. Είμαι σίγουρο ότι ο κύριο Ντόνζο θα επιμείνει σε σχέση με τα θέματα αυτά. Οι γαλλικέ δυνάμει στο Μαλί ετοιμάζουν την αποχώρησή του και ετοιμάζουν να υπάρξει η μετάβαση σε μια δύναμη διατήρηση ειρήνης του ΟΗΕ, αλλά συγχρόνως προετοιμάζεται και η εκλογική διαδικασία στο Μαλί που θα, λάβει χώρα, θα λάβουν χώρα εκλογές τον Ιούλιο και που ελπίζουμε ότι θα νομιμοποιήσουν τις αρχές της χώρας και θα επιτρέψουν στις αρχές αυτές να προχωρήσουν η δικοδόμηση θεσμών στο Μαλί. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Ζολή που είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης στο Κοινοβουλίο μας και μετά μια σειρά από συναδέλφους αλλά ζητώντα σα να προσπαθήσετε πραγματικά να παραμείνετε μέσα στο όριο των δύο λεπτών, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Κύριε Ζωλή, έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τον κύριο Πρόντι που ήρθε εδώ για να μοιραστεί μαζί μας τις σκέψεις του. Όπως ξέρουν όλοι, η κρίση του Μαλή είναι πολύπλοκη και απαιτεί μια συνολική και συνεκτική λύση για να εξασφαλίσουμε μόνιμη ειρήνη. Μετά από το, τα δραματικά γεγονότα και το στρατιωτικό πραξικόπημα του Μαρτίου, οι αρχές του οι αρχές του Μαλή έχουν ανακτήσει ένα μεγάλο μέρος του εδάφους μετά από την ανάπτυξη των γαλλικών στρατευμάτων που υποστηρίζονται από την ε, δύναμη του ΟΗΕ η οποία εκπαιδεύει και τις τοπικές δυνάμεις. Η κατάσταση το βέβαια παραμένει σε εύθραυστο επίπεδο. Το Φεβρουάριο του 2013 έλαβε χώρα μια συνδιάσκεψη για το Μάλι με στόχο να αντιμετωπίσει το θέμα της ανοικοδόμησης του Μάλι με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να αναλάβουν οι ίδιοι οι Μαλιανοί το θέμα της ε, οικοδόμησης της ειρήνης και της ανοικοδόμησης της χώρας τους και να μπορέσουν να συμμετάσχουν πλήρως στην πολιτική και οικονομική ζωή της χώρας τους. Με ποιο τρόπο τώρα η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσαρμόζεται στην ε, κατάσταση που προκέκυψε μετά από τη γαλλική παρέμβαση και πώς προσανατολίζεται στην υποστήριξη της πολιτικής οικοδόμησης θεσμών και την ε, εφαρμογή του οδικού χάρτη. Πώς βλέπετε να λάβει χώρα η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από την απόσυρση των γαλλικών στρατευμάτων, θα εξασφαλίσουμε ότι η ανάπτυξη, η ασφάλεια και η καλή διακυβέρνηση θα μπορέσουν να ενισχυθούν για να ενισχυθεί και η κυβέρνηση του Μαλή. Και ποια είναι τα συμπεράσματα τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή την κρίση για το μέλλον ώστε να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη εφαρμογή πολιτικών και να έχουμε ένα καλύτερο συντονισμό της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να επιταχύνουμε τις παρεμβάσεις όταν είναι απαραίτητες. Η ε, αποστολή εκπαίδευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια μεγάλη συμβολή για να ενισχυθεί η ικανότητα του στρατού του Μαλή και ο δημοκρατικός και πολιτικός έλεγχος τους. Τι μπορεί να κάνει όμω περαιτέρω η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχύσει την μεταρρύθμιση στον ευρύτερο τομέα ασφαλεία και να εξασφαλίσει πολιτική και κοινοβουλευτική εποπτεία των δυνάμεων ασφαλείας στο Μαλί, ώστε αυτές οι δυνάμεις ασφαλείας δεν θα υπονομεύσουν την πορεία προς την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Και τέλος, ποια είναι τα μέτρα με τα οποία θα εξασφαλίσουμε διάλογο στα πλαίσια της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου και Συμφιλίωσης για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια μόνιμη ειρήνη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ντανζάν, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Υποεπιτροπής για τα θέματα ασφαλείας και ο οποίος ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας μας που γύρισε μόλις το Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόντι, σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας η οποία επιβεβαιώνει και τη δική μας διαπίστωση από την αποστολή που κάναμε στο Μαλί και τον Ήγηρα. Αυτό το οποίο μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα στο Μαλί είναι ότι είναι τεράστιος ο κίνδυνος ο οποίος ελοχεύει, ότι οι στατιωτικέ επιτυχίες οι οποίες είναι αδιαφυσβήτητες και οι οποίες επετέθηκαν, να μην μας, θα είναι λάθος να μας δώσουν την εντύπωση αυτές οι, οι επιτυχίες ότι επαρκούν γιατί είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε μια πολιτική διαδικασία διαλόγου και οικοδομηση τη ειρήνης, η οποία πρέπει να αντιμετωπίσει και την προηγούμενη κατάρρευση των θεσμών στο Μαλί. Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό να δει κανεί ότι έχει στον Παμάκο συνομιλητέ που είναι ατομικά απόλυτα αξιόλογοι αλλά δεν έχουν καμία θεσμική βάση και καμία, κανένα θεσμικό ρόλο μέσα στην χώρα αυτή. Το κενό αυτό λοιπόν είναι ηλικιώδες όταν σκέφτεται κανείς τι πρέπει να επιτευχθεί σε οικονομικό επίπεδο, σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο εκλογικών διαδικασιών όπως αναφέρθηκε. Και επομένω ο φόβος μας <clears throat> και το ερώτημα με το οποίο γυρίσαμε από το Μαλί είναι κατά πόσο υπάρχει και μια αντιστοιχία μεταξύ των χρονοδιαγραμμάτων σε διάφορα επίπεδα. Εγώ κατανοώ ότι η Γαλλία επιθυμεί να επαναπατρίσει το ταχύτερο δυνατό τις στρατιωτικές της δυνάμεις, τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος της. Δεν πρόκειται η Γαλλία να αναλάβει όλο το έργο της σταθεροποίησης της χώρας αυτής στο μέλλον, αλλά το, για να μπορέσει να συμπέσει αυτή η ταχεία απόσυση με την ταχεία διοργάνωση εκλογών και την εκκίνηση ενός εθνικού διαλόγου, ο οποίος ήταν πολύ πολύπλοκος και πολυεπίπεδος, αυτά με δυσκολεύουν κάπως να τα κατανοήσω. Βλέπω ότι αυτή η χρονική σύμπτωση περιέχει πολύ, περιέχει πολύ περισσότερους κινδύνους παρά θετικά στοιχεία. Και επίσης ενοχλούμε από το γεγονός ότι βλέπω να υπάρχει μια κάποια σύγχυση μεταξύ όλων αυτών που δρούν επιτοπίους. Έχουμε κάπου 15 ειδικού ε, ε, απεσταλμένους του ΟΗΕ, της Αφρικανικής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, των διαφόρων διοικητών δυνάμεων των τμήματων των στρατιωτικών από τις αφρικανικές χώρες που είναι εκεί, νομίζω ότι αυτά μας οδηγούν σε μια μεγάλη σύγχυση και έλλειψη αποτελεσματικού συντονισμού και στην πρωτεύουσα στον Παμάκο και επί επιτοπίως. Προφανώς λοιπόν όλα αυτά που βλέπουμε μας οδηγούν σε ένα μήνυμα ελπίδας, αλλά συγχρόνως γυρίσαμε και με περισσότερες ανησυχίες από ό,τι είχαμε προτού μεταβούμε επιτόπου στο Μαλί. Θα ήθελα να έχω λοιπόν τη δική σας άποψη για το θέμα του συγχρονισμού των χρονοδιαγραμμάτων που συμπεριλαμβάνει και πολλούς κινδύνους. Χρειάζεται μια μεγαλύτερη θελησιοκρατία σε ό,τι αφορά την ε, πρόοδο προς τις εκλογές και την οικοδόμηση των θεσμών στο Μαλί, αλλά συγχρόνως αυτό πρέπει να συνοδεύεται και από κάποιο ρεαλισμό και κάποια σοφροσύνη για να μπορέσουμε να είμαστε επιτυχείς. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Για δύο λεπτά έχει λόγο. Κύριε Πρόεδρε, να σας ρωτήσω το εξής. Τι ζητάτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην παρούσα φάση. Αξιολογείτε, φαντάζομαι, το τι γίνεται και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ηγηθεί αυτή τη τεράστια ε, προσπάθεια στην περιοχή. Αλλά πείτε μας, γιατί μπορεί να σας βοηθήσουμε, όπως ξέρετε. για να διασφαλίσουμε ότι πραγματικά η Ευρώπη συμβάλλει αυτά που χρειάζεται. Και δεν μιλάω μόνο για χρήματα, μιλάω και για προσωπικό, με τις κατάλληλες ικανότητες για την ανάπτυξη των πολιτικών καθηκόντων που έχετε υπόψη σας. Πώς αξιολογείτε λοιπόν την κατάσταση στο Μαλί και στη γενικότερη περιοχή σε ό,τι αφορά και τις συγκρούσεις στην περιοχή. Δεν μπορούμε φυσικά να μην λάβουμε υπόψη τι γίνεται σε όλη την περιοχή του Σαχέλ. Φυσικά υπάρχει σύνδεση με τη Λιβύη. Και σε ό,τι αφορά την κατάσταση μετά το κατάφη. Υπάρχει σχέση με το πραξικόπημα που είδαμε στην Κεντρική Αφρικανική ε, δημοκρατία. Υπάρχουν φυσικά κίνδυνοι και στον Ήγυρα, Στη Γουινέα Μπισάου, η κατάσταση με το οργανωμένο έγκλημα, τα καρτέλ ναρκωτικών και οι άλλες συγκρούσεις στην περιοχή, ειδικά στη Δυτική Σαχάρα. Πώς θεωρείτε λοιπόν ότι όλα αυτά θα επηρεάσουν την κατάσταση του Σαχέλ. Ευχαριστώ πολύ και θα πρέπει πριν δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή να πω ότι θα αναγκαστούμε να κλείσουμε τον κατάλογο των ομιλητών. Ο κύριος Μπούζεκ έχει το λόγο και είναι τελευταίος, γιατί θα πρέπει να δώσουμε το λόγο στον ε, κύριο Πρώτη για να απαντήσει. Ο κύριος Βάικελ είναι επόμενος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας βλέπουμε εδώ. Νομίζω ότι εσείς είστε το κατάλληλο άτομο που μπορεί σε αυτή την περιοχή που δοκιμάζεται από τόσα πολλά προβλήματα μπορείτε να εδραιώσετε μια προσέγγιση η οποία να είναι εξισορροπημένη. Και τώρα θα μιλήσω στο σλοβένικα. Συμφωνώ μαζί σας. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ μαζί σας ότι η περιοχή αυτή ε, επιβαρύνεται από καινούργια αλλά και από παλιά προβλήματα. Έχουν διαμορφωθεί ε, νέε καταστάσει, νέα προβλήματα, τα οποία δύσκολα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί. Αλλά θα ήθελα να επισημάνω και ένα παλαιό πρόβλημα, το οποίο το επισήμανε και η συνάδελφο Γκόμε. Και μάλιστα επειδή η κατάσταση αυτή επηρεάζει και τα γενικότερα προβλήματα. Ε, φυσικά στο πρόβλημα της Δυτικής Σαχάρας. Η κυβέρνηση του Μαρόκο πριν από κάποιο καιρό ανακοίνωσε ότι διώχνει μία σειρά εντεταλμένων της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης που ήθελαν να επισκεφτούν τη Δυτική Σαχάρα προκειμένου να διαπιστώσουν κατά πόσο υπάρχουν, ε, τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα μια ομάδα ευρωβουλευτών. Και το θέμα λοιπόν τώρα είναι κύριε Πρόντι, κατά πόσον εσείς θα καταβάλλετε προσπάθειες προκειμένου η αντιπροσωπεία της ε, Ινούσο θα λάβει εντολή. προκειμένου να παρακολουθήσει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δυτική Σαχάρα. Ιδάλω θα επιδεινωθεί περαιτέρω το θέμα και το πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ματού. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για τον κύριο Πρόεδρε έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά το θέμα των Τουαρέγ. Οι Τουαρέγ είναι ομάδες. Δεν είναι μόνο στο Μαλί. Ε, πώς βλέπετε την κατάσταση, ότι υπάρχουν εθνικιστικές τριβές Πώς βλέπετε την επιβίωση των Τουαρέγ σε αυτή την περιοχή. Και το δεύτερο ερώτημα αφορά το σημαντικό ρόλο που παίζει η διασπορά του Μαλή στην Ευρώπη και κυρίως στην Γαλλία. Πώς βλέπετε τη συνεισφορά τους, γνωρίζοντας ότι ήδη η διασπορά του Μαλή χρηματοδοτεί τους πληθυσμούς που ζουν στο Μαλή ε, πώς θα τους εντάξετε αυτούς στον όλο προβληματισμό και στη δράση που θέλετε να εφαρμόσετε στο Σαχέλ και στο Μαλί πιο συγκεκριμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Τσάρλς Τάνοκ. Α, πρόεδρε. Εδώ είμαι κύριε πρόεδρε. Είμαι συγκητής του Κοινοβουλίου για μια έκθεση που δεν έχει συνταχθεί ακόμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Σαχέλ που θα συμπεραβάνει και τη Δυτική Σαχάρα που θα είναι τεράστια πρόκληση όπως και τα στρατόπεδα στην Αλγερία, οι στην Αλγερία και θα εξεταστούν όχι μόνο θέματα αμήνης και ασφαλείας έναντι του Μαλή, αλλά και θέματα όπως η καζόμενη δουλεία που εφαρμόζεται στη Μαυριτανία, η ομοίη εφαρμογή του Σαρία ε, στον Βόρειο Μάλι, το θέμα του εμπορίου ανθρώπων που δυστυχώς συνδέεται με το λαθρεμπόριο όπλων και ναρκωτικών σε, μια λεωφόρο που ξεκινά από τη δυτική ακτή της Γουινέας Βυσάου και την Ιγυρία και πάει στο Μπόκο Χοράμ και περνάει από όλο το Σαχέλ και πάει στις ομάδες Al-Shabaab, στην ομάδα Shabaab στη Σαμαλία. Πρώτη ερώτηση, ποιος ο ρόλος, αν υπάρχει ρόλος για φιλικές χώρες όπως είναι το Κατάρ, που εξακολουθούν να εξοπλίζουν οι Ισλαμιστές. Ε, ξέρουμε ότι υπάρχει υπερχείληση από τη Λιβύη, ίσως να υπάρχει ροή όμως όπλων και από χώρες όπως είναι το Κατάρ. Η ερώτησή μου, τι μπορεί να γίνει για να λυθούν τα προβλήματα των του Οπότε το MNLA ε, έχει μετακινηθεί. Ε, οι Ισλαμιστές έχουν μετακινηθεί λόγω γαλλικής παρέμβασης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πώς μπορεί να εκπαιδεύσει τις δυνάμεις του Μαλή και τις δυνάμεις των Ήγυρα. Υπάρχει κίνδυνος για τα, να πέσει στα χέρια των τζιχαντιστών στον Ήγυρα τα ορυχεία του ουρανίου και να κατασκευάσουν μικροπυρηνικές βόμβες που μπορούν να απειλήσουν τους πολίτες μας. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κράτο στην περιοχή. Υπάρχει κρίση στην Ευρωζώνη, μπορούμε να μάθουμε τίποτα από αυτή την περιοχή. Διότι φαίνεται ότι είχαν πολύ το κοινό νόμισμα, κοινό αφρικανικό φράγκο επί χρόνια που συνδεόταν με το ευρώ. Πώ μπορεί να το καταφέρουν αυτό και δεν μπόρεσε να καταφέρει κάτι τέτοιο η Ευρωζώνη. Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Και τώρα να καλέσω τους προέδρους των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων από την Αλγερία, το Μαρόκο και την Τινησία να τους ρωτήσουν θέλουν να μιλήσουν. Θα αντιμετωπιστούν ισότιμα. Δύο λεπτά έχουν ο καθένας αν επιθυμούν να παρέμβουν. Ο κ. Μπελκασέμ, αν επιθυμεί, μπορεί να ξεκινήσει. Ας ακολουθήσουμε μια αλφαβητική ε, σειρά, λοιπόν. Πατήστε το κουμπάκι σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι πολύ ευτυχής για την πρόσκληση που μας απευθύνατε, που μας επίφθινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συζητήσουμε το κρίσιμο πρόβλημα της περιοχής του Σαχέλ. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Πρόντι, ο οποίος ήδη άρχισε να αναφέρεται στο θέμα, πολύ δύσκολο, αλλά θα πρέπει να μπούμε και στο αίτιο. Για την αποσταθεροποίηση του Μαλή είναι κοινωνικά τέτοια την αποσταθεροποίηση και τρομοκρατία. Η τρομοκρατία που εδρεύεται στην περιοχή του Σαχέλ που υπονόμευσε αυτή τη χώρα, η τρομοκρατία και αυτή η τρομοκρατία τώρα ε, για να πετύχουν σταθεροποίηση πρέπει να κρυζωθεί η τρομοκρατία. Για να εκριζώσουμε λοιπόν την τρομοκρατία από την περιοχή θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τη χρηματοδότηση των τρομοκρατών η τρομοκρατία και η χρηματοδότηση τρομοκρατίας προέρχεται από το εμπόριο όπλων, από τα λίτρα και από το εμπόριο ναρκωτικών. Ε, το ναρκωτικό έχει μεγάλη θέση σε αυτή τη λωρίδα του Σαχέλ ε, και θα πρέπει αυτό να, να σκεφτούμε αυτή τη μάστιγα που πλήττει πάρα πολλές χώρες. Και η χώρα μου πρόσφατα μπόρεσε να θέσει τέρμα σε ένα εμπόριο ε, το 2012 για 100, που ήταν 157 τόνοι χασίς που κατασχέθηκαν στα σύνορα. Η πηγή της χρηματοδότησης πιστεύω των τρομοκρατών πρέπει να καταπολεμηθεί. Να καταπολεμηθεί η χρηματοδότηση. Κύριε Πρόντι, συμμερίζομαι ε, μαζί σας την άποψη πρέπει να συνδυαστούν οι προσπάθειες, οι αναπτυξιακές και οι προσπάθειες για την ασφάλεια. Άρα πρέπει να δραστηριοποιηθεί η διαδικασία του 2011, η διάσκεψη υψηλού επίπεδου ε, συνεργασίας ασφάλειας και ανάπτυξης. Είμαστε έτοιμοι να διοργανώσουμε το Αλγέρι 2, γιατί αυτό ήταν το Αλγέρι 1, για να ενεργοποιηθεί όλη η δραστηριότητα αυτή τη σύμπραξη για την ασφάλεια, και την ανάπτυξη στην ε, περιοχή. Κύριε Πρόντι, όπως είπατε πολύ καλά, όπως και πολλοί ευρωβουλευτές και συμφωνώ μαζί τους είπαν, αυτή η περιοχή ακόμα αντιμετωπίζει σοβαρές ε, δυσκολίες όσον αφορά την ασφάλεια. Τα προβλήματα δεν έχουν διευθυνθεί και βλέπετε ότι η τρομοκρατία ε, έχει διαστάσεις διεθνείς. Έχει δεχθεί επιθέσεις από διεθνή ομάδα τρομοκρατική χώρα μου, η οποία είχε σαν στόχο μία βάση, μία μονάδα υγροποίησης ε, φυσικού αερίου Τελευταία έγινε αυτή η επίθεση και ευτυχώ η Αλγερία επομίστηκε τι ευθύνε τη και δεν επέτρεψε σε αυτού του τρομοκράτε, την ομάδα των τρομοκρατών, να κρατήσει τους ομήρου. Να πάρει τους ομήρου και να τους μεταφέρει προς το Μαλί και να του χρησιμοποιήσει σαν ε, ομήρου για εκβιασμούς. Λοιπόν, χρειάζεται λοιπόν η προσέγγιση από την ασφάλεια και έχουμε ένα έγγραφο το οποίο με τίτλο «Συμπερόσματα της Νουαξότ» που ήταν αντικείμενο συζητήσεων από όλες τις χώρες της περιοχής. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μια βάση για τις συζητήσεις ε, και για προβληματισμό. Τώρα, όσον αφορά την πολιτική λύση. Η Αλγερία πάντα ήταν υπέρ της πολιτικής ε, λύσεως για το πρόβλημα του Μαλή, όμως ε, θα πρέπει να υπάρξει μια προσέγγιση ε, χωρίς να υπάρχουν αποκλεισμοί. Δεν πρέπει κανείς να αποκλειστεί από το διάλογο και νομίζω ότι για να υποστηρίξουμε τις προσπάθειές σας, όπως είπε και ένας συνάδελφος ευρωβουλευτής, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πολλές αποστολές. Πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τις, τα έργα των αποστολών. Πώς μπορούμε στο μέλλον, κύριε Πρώτη, να ε, συντονίσουμε το έργο των αποστολών. Θα πρέπει, όπως είπε και κάποιος ε, ευρωβουλευτής, να όλοι οι και η διασπορά να συμμετάσχει στην προσπάθεια των χωρών. Να δημιουργηθεί μια επιτροπή σοφών στη διασπορά που να μπορεί να βοηθήσει στη διευθέτηση των προβλημάτων και την εξέβρεση λύση. Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό μαλλί που να μπορεί το μαλλί να λύσει τα δικά του προβλήματα μόνο του. Χρειάζονται βιώσιμες λύσεις για να μπορέσουμε να δώσουμε σε αυτή τη χώρα ελπίδα, ε, ελπίδα στο λαό του Μαλή. Ευχαριστώ. Ο κύριος έχει το λόγο. Του Μαρόκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χωρίς μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μαρίκ Περί, Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Μαροκινού Κοινοβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε η επισταλμένε το, του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ, αγαπητοί ευρωβουλευτές, θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μας απευθύνατε προς το Μαροκινό Κοινοβούλιο, ώστε να σας παρουσιάσω τις θέσεις μας για τα θέματα αυτά που έχουν να κάνουν με την κατάσταση στη Σαχάρα και στο Σαχέλ. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα επίκαιρη αυτή η συνεδρίαση και έχει ε, λάβει χώρα σε ένα ε, συγκεκριμένο πλαίσιο για, για λόγους που είναι πολύ σημαντικοί. Πρώτα απ' όλα έχουμε την ε, σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή μας. Μια έκθυλη επιδείνωση ασφαλείας σε μια περιοχή την οποία ο κύριος Πρόντι ανέφερε ότι έχει ένα μήκος 5.000 χιλιόμετρων και πλάτος 1.000 χιλιόμετρων. Πρόκειται λοιπόν για μια απειλή και γεωγραφικού χαρακτήρα η οποία εκτείνεται σε τεράστιες αποστάσεις που ποτέ δεν είχαν παρουσιαστεί στο παρελθόν στις προηγούμενες συγκρούσεις. Ένας δεύτερος λόγος έχουμε τον πολλαπλασιασμό των απειλών. Υπάρχει τρομοκρατική απειλή, υπάρχει το τεράστιο λαθρεμπόριο όπλων που λαμβάνει η χώρα, το τεράστιες έκταση λαθρεμπόριο ναρκωτικών που εμπλέκει και χώρες Λατινικής Αμερικής και που διαμετακομίζονται τα ναρκωτικά από τις περιοχές αυτές μέχρι ότου φτάσουν κυρίως στην Ευρώπη και φυσικά υπάρχει και το θέμα της λαθρεμπορίας ανθρώπων και οι παράνομες μεταναστευτικές ροές. Τρίτον, έχουμε ένα πολλαπλασιασμό των εμπλεκομένων. Υπάρχει η Al-Shabaab, όχι μόνο η Al-Qaeda, υπάρχει η Boko Haram και άλλοι οργανισμοί που ασκούν την τρομοκρατία. Το Μαρόκο έχει ήδη κρούσει τον κόντρο του κινδύνου σε σχέση με την κατάσταση στην περιοχή αυτή εδώ και πολλά χρόνια και σε το πιο υψηλό επίπεδο, σε επίπεδο αρχηγών κρατών, ο Αχπετοέκτος, ο βασιλεύς του Μαρόκου, στις 31 Ιουλίου 2010, στην ομιλία που έκανε κατά την ενθρόνησή του, αναφέρθηκε σε αυτή την τρομοκρατική απειλή. Δυστυχώ, δεν έτειναν ευήκον ους οι λήπτες αποφάσεων σε άλλους χώρους. Για το Μαρόκο, για την εδαφική ακαιρεότητα της χώρας μας. Η αποσχιστική κίνηση η οποία έχει δημιουργηθεί στο Βόρειο Μαλή είναι μία απειλή και εμείς έχουμε τονίσει τη θέση μας για την διατήρηση εδαφικής ακαιρεότητας του Μαλί. Η Γαλλία, της οποίας εδώ χαιρετίζουμε το θάρρος, διότι ανέλαβε μία στρατιωτική ενέργεια η οποία ε, νομοποιήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας με τις χώρες της Δυτικής Αφρικής και το Μαρόκο που την υποστήριξαν έχει κάνει τεράστια προσπάθεια και έχει κρατήσει το Μαλί εν ζωή γιατί αλλιώς θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ πιο <clears throat> δραματική κατάσταση. Το Μαρόκο συμμετέσχει επίσης και σε ανθρωπιστικό επίπεδο στη βοήθεια που δόθηκε στους πρόσφυγες από το Μαλί οι οποίοι μετακινήθηκαν σε άλλες χώρες. Και έχει επίσης συμμετάσχει το Μαρόκο με χρηματοδότηση 5 εκατομμυρίων δολαρίων για τις δυνάμεις της Ένωσης της Δυτικής Αφρικής. Ποια είναι τώρα η απάντηση πρέπει να δοθεί σε αυτή την κατάσταση. Ένα κράτος μόνο του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Χρειάζεται να υπάρξει συντονισμός των προσπαθειών όλων των χωρών της περιοχής. Πρέπει να υπάρξει και συνεργασία με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οι πολίτες της πολλές φορές είναι ο προνομιακός στόχος αυτών των τρομοκρατών. Δεύτερον, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η περιφερειακή ολοκλήρωση των χωρών του Μαγκρέπ δεν είναι μονάχα θέμα οικονομικό αλλά και θέμα ασφάλειας. Και τέλος τονίζω ότι η συμμετοχή μιας χώρας, μιας μικρής ομάδας χωρών στην περιοχή δεν είναι επαρκής και το Μαρόκο είναι απόλυτα διατεθειμένο να θέσει την εμπειρία του στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας. Ευχαριστώ που μας καλέσατε να παραστούμε σε αυτή την συνεδρίαση. Ευχαριστώ λοιπόν που μας υποδεχθήκατε στο Κοινοβούλιο και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που προσδίδετε στα ανθρωπιστικά ζητήματα. Βέβαια, το πραξικόπημα στο Μαλί τον Μάρτιο συνέβαλε κατά πολύ στην ενίσχυση της τρομοκρατίας στην περιοχή του Σαχέλ. Αυτή η τρομοκρατία δεν μπορεί να απομονωθεί σε μια χώρα. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, δεν υπάρχουν σύνορα για την τρομοκρατία. Δεν γνωρίζει σύνορα η τρομοκρατία. Η τρομοκρατία είναι το παρόν πρόβλημα. Και αυτή η τρομοκρατία δεν οφείλεται σε ιδεολογικά ζητήματα. Αλλά η τρομοκρατία είναι συνέπεια μιας κρίσεως, μιας μεγάλης κρίσεως που οφείλεται στο εμπόριο ε, ναρκωτικών και το εμπόριο ανθρώπων. Αυτή είναι η πηγή αυτή είναι η βάση της τρομοκρατίας στην περιοχή. Η παρούσα κατάσταση είναι ευαίσθητη στο Μαλί. Δεν εξαιρούνται από τα προβλήματα οι γειτονικές χώρες, όπως η Αλγερία, που είναι πολύ κοντά στην Τινησία και κοντά στην ε, Λιβύη. Αυτή η τρομοκρατία, αυτού του είδους η τρομοκρατία, ε, ε, ξεκίνησε και ενισχύθηκε και μετά την ε, Αραβική Άνοιξη. Με το κάποιο τρόπο συνέβαλε στην αλλαγή και στο εμπόριο όπλων. Μετά από αυτά που έγιναν στη Λιβύη αυξήθηκε το εμπόριο όπλων και αυτό συνέβαλε κατά πολύ στη διαφθορά και συνέβαλε και στην τρομοκρατία και την εδραίωση της τρομοκρατίας στην περιοχή. Εμείς στην Ισία καταδικάζουμε την βία και την τρομοκρατία και τον διαχωρισμό, τον διαμελισμό της χώρας και εκφράζουμε ανησυχία όσον αφορά την ανασφάλεια που επικρατεί στο Μαλί και την επιδείνωση της ανθρωπιστικής καταστάσεως, κυρίως στο βόρειο τμήμα της χώρας και επιμένουμε επί της σημασίας της εδαφικής ακαιρεότητας του Μαλί και καταδικάζουμε κάθε απειλή που ε, προέρχεται από τις ένοπλες τρομοκρατικές ομάδες. Κατανοούμε τη γαλλική απόφαση και την ευρωπαϊκή απόφαση που αφορούν την ανάγκη που υπάρχει για την επίλυση των προβλημάτων και μετά από την πρωτοβουλία της Γαλλίας και την απόφαση απόσυρσης των γαλλικών δυνάμεων από το Μαλί καταλάβαμε τις αποφάσεις που ελήφθησαν και θεωρούμε ότι μια πολιτική ε, βούληση, πραγματική πολιτική βούληση είναι πάρα πολύ σημαντική για να βρεθεί κάποια λύση και για να μην καταστραφεί ο λαός ε, χρειάζεται να, να εξεταστεί το θέμα Χρειάζεται μια πρωτοβουλία με διεθνή νομιμότητα. Χρειάζεται μια επιχείρηση σταθερότητας που θα επιτρέψει την οικονομική ανάπτυξη και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πιστεύω ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να έχουν πολύ θετικά αποτελέσματα στην περιοχή, αν επιτευχθούν. Θα ήθελα να επιμείνω επίσης και επί Η Τινησία στη συνεδρίαση των δωρητών δεσμεύτηκε να χρηματοδοτήσει την ανοικοδόμηση του Μαλή, να συνδράμει και στην, ανικοδό στην ανόρθωση του στρατού και στην εκπαίδευση σε πολυμερές επίπεδο του στρατού. Σε επίπεδο πολιτικό υποστηρίζουμε την διοργάνωση εκλογών το ταχύτερων δυνατών. Ε, πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε ειρηνική λύση, να επεξεργαστούμε μια στρατηγική, ένα σχέδιο εργασίας σαφές, που θα επιτρέπει να περάσουμε από μια προβληματική κατάσταση σε μια κατάσταση πιο σταθερή και πιο λογική, πιο, πιο ευνοϊκή για την ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Okay. Ευχαριστώ που είστε εδώ, Πρόεδρε Πρόντι, λέει ο κ ε, σας έθεσα να ρωτήσω για τον ρόλο του ΟΗΕ. Εγώ έχω κάποιες παρατηρήσεις να θέσω για να δω πώς βλέπετε από πολιτική σκοπιά τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση που θέλω να σας θέσω είναι η εξής. Αν μια ιδιαίτερη πολιτική ασφαλείας που εγγενιάστηκε σε αυτή την περιοχή μετά το 2001 μετά την επίθεση του δίδυμου πύργου, αν αυτή η πολιτική δεν έδωσε κίνητρα σε μια, δεν οδήγησε σε μια οικονομική κοινωνική ε, φτώχεια που είναι στη ρίζα των προβλημάτων. Δεύτερη ερώτηση που εν μέρη ετέθη και από την Άννα Γκόμε. Πώς επηρέασαν τα γεγονότα στη Λιβύη τα προβλήματα που ήδη υπήρχαν στο Βόρειο Μάλι. Τέλος, συμφωνώ μαζί σας. Πράγματι χρειάζεται μια στρατηγική συντονισμένη και ολοκληρωμένη. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες του ΙΕ θα πρέπει να επικεντρώσουν την προσοχή τους επί τεσσάρων αξώνων που αναφέρω ακροθυγώ για να καταλάβετε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρξει νέα προσέγγιση όσον αφορά την πολιτική γειτονία τη Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πρέπει να είναι διαφορετική σε σχέση με το παρελθόν όπου ε, έγιναν πολλά σφάλματα. Δεύτερη δεύτερος άξονας που αναφέρθηκε από τους εκπροσώπους των τριών χωρών που καλέσαμε εδώ, χρειάζεται μια καλύτερη πολιτική με μεγαλύτερα αποτελέσματα από πλευράς Μαγκρέμπ στην περιοχή για μεγαλύτερη σταθερότητα. Τρίτη πτυχή, τρίτο άξονα που δεν υπογραμμίστηκε, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό άξονα για να εδρεωθεί η δημοκρατία σε αυτή την περιοχή. Ανάπτυξη τη κοινοβουλευτική διάσταση, που είναι μία από τι αποφασιστικέ διαστάσει. Και τέλο, Πιστεύω ότι θα πρέπει μαζί να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε μια, κάποια επικοινωνική προσέγγιση ε, που ακολουθούν κάποια κάτι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν έτσι σχέσεις τέτοιου είδους με τις χώρες περιοχής. Χρειάζεται συνεργασία για να υλοποιήσουμε τους στόχους και θα ήθελα να ξέρω ποιες είναι οι απόψεις για αυτά που σας είπα. Ο κύριος Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να σας συγχαρώ για την διοργάνωση αυτής της ε, συνάντησης και ιδίως για το γεγονός ότι είναι παρόντες και οι πρόεδροι των τριών επιτροπών εξωτερικών των χωρών του Μαγρέπ. Εγώ δεν είχα την ευκαιρία να ακούσω αυτά που είπε ο πρόεδρος Πρόντι γιατί ψήφισα σε μια άλλη επιτροπή. Αλλά θα ήθελα να τον καλωσορίσω εδώ. Είναι φίλος από πολύ παλιά και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να σας θέσω ορισμένα ερωτήματα γιατί σε μια προηγούμενη μετεσάρκωση του ο πρόεδρος ε, Πρόντι ήταν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φίλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Πρόντι πώς η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της κρίσης στο Σαχέλ πέραν των θεμάτων εκπαίδευση που έχει αναφερθεί ήδη, αν θεωρεί ότι είναι επαρκής για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερα επίπεδα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Το δεύτερο ερώτημά μου έχει να κάνει με το κατά πόσο θεωρείται ότι η νέα ε, η ανανεωμένη μεσογειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επαρκής ώστε μέσα από τα διάφορα συστατικά της στοιχεία να προκύψουν δυνατότητες ανάπτυξης για τις χώρες της περιοχής. Και τέλος, όπως είπε και ο κ. Ντανζόν προηγουμένως, θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο ο πρόεδρος πρώτη, πιστεύει ότι η δράση των διαφορέων διαφορετικών φορέων που είναι παρόντες στο χώρο της κρίσης έχουν συμπληρωματικό και συνεκτικό χαρακτήρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βουάτσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να σας πω πόσο σας ευχαριστούμε που κάποιος με τόση εμπειρία, και, όπως ο Ρωμάντο Πρόντι, μπορεί να βρεθεί εδώ πέρα και να εκφράσω τη χαρά μου που βρίσκεστε εδώ. Θα ήθελα να σας θέσω δύο ερωτήσεις, Πρόεδρε. Τι μπορούμε να κάνουμε στην περιοχή του Σαχέλ προκειμένου να βελτιώσουμε την ανάπτυξη δυναμικού για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, δηλαδή για να βελτιωθεί η ικανότητά μας όχι μόνο να συνεργαζόμαστε με τις κυβερνήσεις, αλλά για να δημιουργηθεί και μια κοινωνία των πολιτών, για να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία για τον κίνδυνο αυτό. Και δεν ξέρω κατά πόσο η Ένωση κάνει τίποτα προς την κατεύθυνση αυτή. Και κατά δεύτερον, ένα πολύ πιο ευρύ ερώτημα, για το οποίο δεν υπάρχει κάποια προφανής λύση. Σε, ποια, σε ποιο βαθμό πιστεύει ο Ρωμανό ότι η αλλαγή του κλίματος και ο αντίκτυπος της καθιστά την κατάσταση όλο και πιο δύσκολη. Ευχαριστώ κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόντι, έχω μία ερώτηση στον αφορά το Μάλι. Όπως γνωρίζουμε όλοι, στο Μαλί πολιτική κρίση προηγήθηκε της κρίσης ασφαλείας και της θετικής παρέμβασης. Και τώρα μετά από χθεσική σχετική σταθεροποίηση θέλουμε να διοργανώσουμε και εκλογές. Το ζητά αυτό η Ένωση και ελπίζουμε ότι η Ένωση θα έχει αποστολή παρατηρήσεως των ε, εκλογών. Σε αυτό το πλαίσιο, με ποιο τρόπο θεωρείτε ότι μπορεί, μπορεί να συμμετάσχει ο ΙΕΣ στην εκλογική διαδικασία. Εγώ έχω εμπειρία από μια χώρα σχετικά κοντινή, την ακτή Ελεφανταστού. Ήμουν επικεφαλής αποστολής στην ακτή Ελεφανταστού και εκεί ο ΙΕ αποφάσισε να κυρώσει τις ε, εκλογές. Βασίζεστε, θεωρείτε ότι μπορεί να γίνει με τέτοια πιστοποίηση, αν θέλετε, να γίνει εξακρίβωση, αν γίνονται σωστά εκλογές και αν ναι, πότε θα γίνει, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για να γίνει αυτή η επιτήρηση των εκλογών. Ε, πότε θα γίνει αυτό, θα γίνουν οι εκλογές Ιούλιο-Αύγουστο. Κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε ότι είναι διαφορετική η οπτική μας γωνία για το μαλή Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρότεινε ένα εντυπωσιακό πακέτο και παρήχε εντυπωσιακό πακέτο βοήθειας. Μισό Μισό δισεκατομμύριο για την μακροπρόθεσμη τροπιστική βοήθεια. Η σημερινή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΟΗΕ σε τι επίπεδο βρίσκεται, σε ό,τι αφορά δηλαδή τη διαχείριση του πακέτου αυτού και κατά τα άλλα, τι κάνουν οι άλλοι διεθνείς φορείς για το Μαλί. Ευχαριστώ. In <laughs> Mr. President, the floor is yours. Μιλήσω και αγγλικά αν θέλετε, αλλά όταν ήμουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποτέ δεν μιλούσα Ιταλικά, αλλά στο Κοινοβούλιο πάντα Ιταλικά. αυτή είναι οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Καλώς συνεχίζει Ιταλικά. Ο οποίος πρώτη σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις, ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρονοδιάγραμμα. Δεν είναι εύκολο να απαντήσω στο χρόνο που μου διατίθεται. Θα απαντήσω συνοπτικά, αλλά αρκετά πλήρης είναι οι απαντήσεις μου. Πρώτη σειρά ερωτήσεων ετέθη, ξεκινώντας από τον πρώτο Ευρωβουλευτή, Ζολή, αφορούσε τη γενική θέση δέσμευση ε, της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανέλαβε πολύ μεγάλη υποχρεώση η Ευρωπαϊκή Ένωση Πρώτα απ' όλα τεχνική βοήθεια. Την 1η Απριλίου φέτος, τώρα δηλαδή, ξεκίνησε η απριλιου φετο τωρα δηλαδη ξεκινησε η αποστολη στο Μάλι EUTM ε για το εμπόριο, το trading. Σημαντική αποστολή. 15 μήνες είναι η αποστολή με 300 εκπαιδευτές, trainers. Η ε, από την, από την αρχή του 2012 κινητοποίησε 115 εκατομμύρια ευρώ Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι πολύ σημαντική, χρήσιμη βοήθεια αυτή, διότι το τεράστιο είναι το βάρος των προσφύγων. Μίλησα με τον Κουτιέρες στον ΟΗΕ για το θέμα αυτό και πράγματι η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη διότι προστίθεται αυτή η κατάσταση και σε άλλες, στην κρίση που έχει γενικά κόσμο. Άλλα 338 εκατομμύρια ευρώ δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την κρίση όσον αφορά τα τρόφιμα. Αλλά ήδη δεσμεύτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε 160 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη της περιοχής στο 10ο πρόγραμμα ανάπτυξης. 2007-2013. Αυτό πάγωσε, πάγωσε αυτό, λόγω της επανάστασης, ας το πούμε έτσι, των εντάσεων στο Μαλί, στο εσωτερικό του Μαλί, πάγωσε αυτή η βοήθεια. Θα επανεργοποιηθεί, πιστεύω, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή η βοήθεια θα επανενεργοποιηθεί όταν ομολοποιηθεί η κατάσταση. Υπάρχει νέο εκπρόσωπος, ε, ο Ευρωπαίος εκεί που πιστεύω ότι θα μπορέσει να συμβάσει την προσπάθεια και υπάρχει και μια διάσκεψη 15 Μαΐου εδώ στις Βρυξέλλες που προβλέπεται να γίνει για το Μαλί. Όχι Σαχέλ, αλλά ήδη υπάρχει σχετικό συντονισμός. Διότι άκουσα και αυτό που είπατε. Να προσέξουμε Αυτό που αισθάνομαι και εγώ. Ο μεγάλος πολυσχηδής επιμερισμός των ευθυνών οδηγεί σε δυσκολία συντονισμών. Δυσκολία συντονισμού και είναι πρωταρχικό πρόβλημα. Και εγώ σαν εκπρόσωπος του ΟΗΕ στο Σαχέλ προσπαθώ να μην ξεφύγω από το σαφέστα το πλαίσιο που έχω, την εντολή που έχω, να συνεργαστώ με τους άλλους υπευθύνους σε στενή επαφή πάντα, όχι μόνο με τους συναδέλφους που έχουν ειδικέ ευθύνες για διάφορους τομείς στον ΟΗΕ, αλλά με ειδικού απεσταλμένους της Αφρικής, είμαστε σε επαφή μαζί τους, με την Αφρικανική Ένωση, είμαστε σε συνεχή επαφή και με όλους τους άλλους εκπροσώπους, ούτω ώστε να μην δημιουργήσουμε σύγχυση, αλλά ενότητα στη δράση. Ε, και αυτό είναι σημαντικότατο και πιστεύω ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ευθύνη, ιδιαίτερη ευθύνη στο ζήτημα αυτό. Συντονισμός λοιπόν έχει μεγάλη σημασία. Αλλά αυτό θα πρέπει να το εντάξουμε κάπου. Πολλές ερωτήσεις αναφέρθηκαν σε αυτό. Χρειάζεται αυτός ο διάλογος της συμφιλίωσης πολύ γρήγορα να γίνει εντός μαλλί. Χωρίς αυτό το διάλογο και η διεξαγωγή των εκλογών κινδυνεύει. Εγώ δεν συμφωνούσα για τις γρήγορες εκλογές πριν τη γαλλική δράση, διότι πολλά τμήματα της χώρας ήταν εκτός. Δεν μπορεί να διοργανώσει κανείς εκλογές που ουσιαστικά θα είχαν διαιρέσει περισσότερο τη χώρα. Τώρα αυτό είναι εφικτό και υποχρεούμεθα να κινηθούμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Δεν είναι εύκολο αυτό. Εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπιστέντα άτομα υπάρχουν που έπρεπε να, να φύγουν, να το σκάσουν από το σπίτι τους. Και έχουμε και το πρόβλημα των εκλογικών καταλόγων, το πρόβλημα. Και αυτές τις ημέρες αυτό αντιμετωπίζεται. Πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει ό,τι γίνεται για να γίνουν τον Ιούλιο πράγματι οι εκλογές. Δεν σας κρύβω τη δυσκολία που αντιμετωπίζει αυτή η διαδικασία και τις μετεωρολογικές δυσκολίες που συνήθως δημιουργούνται τον Ιούλιο διότι εκείνο το μήνα είναι ε, πολύ δύσκολες συνθήκες. Εάν όμως δεν ξεκινήσουμε με γρήγορους ρυθμούς, δεν θα γίνουν εκλογές. Και ξέρω πολύ καλά, θυμηθείτε το, ότι αν δεν περάσουμε από εκλογική διαδικασία το πρόβλημα του Μαλή είναι ανεπίλητο, διότι οι εσωτερικές εντάσεις, οι συγκρούσεις που έγιναν μετά το πραξικόπημα, ο διχασμός ιδιαίτερης εξουσίας είναι τέτοια στοιχεία, χωρίς να ξεφύγει κανείς από τη διαδικασία μέσω εκλογών, δεν μπορούμε να έχουμε ένα μάλι το οποίο θα είναι αποτελεσματικό και πραγματικά μπορεί να κινηθεί προς το μέλλον. Δεν είναι ρητορικό σχήμα οι εκλογές. Σε αυτή την περίπτωση οι εκλογές δεν είναι μόνο η αρχή δημοκρατικής διαδικασίας. Είναι ένα σπάσιμο με το παρελθόν. Ξεφεύγει η χώρα από το παρελθόν. Αλλιώς θα μπορούσε συνεχιστεί η κατάσταση ένα, Διότι αυτούς τους μήνες εγώ προσπάθησα Είδα τι έγινε με την απονομή των ευθυνών, τα παιχνίδια που γινόταν εδώ στις χώρες, τα προβλήματα που υπήρχαν να ακούσει κανείς μια ενιαία τοποθέτηση για να καταλάβει τι συμβαίνει. Εγώ υποστήριξα πάρα πολύ το ότι οι κυβερνώντες τώρα βγήκαν εκτός της πολιτικής μάχης, αφήνοντας ένα πιο ελεύθερο μέλλον για τη χώρα. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο και σημαντικό. Έτσι δε περαιτέρω διότι είναι σημαντικέ και εκλογέ. Και πιο σημαντικέ είναι οι εκλογέ σε αυτή την περίπτωση. Διότι έτσι σπάμε από το, την κατάσταση εξόδου. Αλλάζουμε ριζικά, ριζική αλλαγή. Διαφορετικά θα ήταν η αλλαγή. Τώρα πιστεύω σε κάτι άλλο. Το να ξεκινήσουν οι διαπραγματευτικέ διαδικασίε αμέσω. Διαφορετικά ε, είναι σαφές ότι υπάρχουν συμφέρει την κυβέρνηση του Μαλή να μείνουν οι Γάλλοι στις θέσεις τους και να κοιμηθεί ούτως η η κυβέρνηση και να, να αναβάλει τις λύσεις. Η διεθνής κοινότητα έχει καθήκον να επιμείνει μέχρι σότου, μέχρι της ανέδειας, να πιέσει, να πιέσει πολύ για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Να γίνουν οι συνομιλίες συμφιλίωσης, να ξεκινήσει ο διάλογος με το Βορρά, να γίνουν οι συνομιλίε που πρέπει να γίνουν. Διότι είναι σαφέ ότι δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την ιστορία του παρελθόντο. Ποιο ήταν το παρελθόν. Συμφωνίε κακοργανωμένε που δεν τηρήθησαν. Συνεπώ υπάρχει καχυποψία και ένταση πολύ πιο μεγάλη από, να από αυτή που μπορούσα να φανταστώ πριν ξεκινήσω αυτή τη δουλειά που κάνω. Είναι σαφές λοιπόν ότι από αυτή την έποψη απαντώ στον κύριο Ντανζάν λέγοντας ότι προφανώς το πρόβλημα της απόσυνσης των γαλλικών στατευμάτων μπορεί να είναι ένα πρόβλημα σταδιακό να αποφασιστεί από τη Γαλλία να γίνει σταδιακά, αλλά θα πρέπει να λάβει υπόψη και την ανάγκη που υπάρχει πάντα που να μπορεί να το χειριστεί το πρόβλημα αφρικανικός κόσμος στο βαθμό τον, τον εφικτό και πιο γρήγορα, με βοήθεια απ' έξω. Αλλά μία απόσυση των στρατευμάτων που θα γίνει τέτοιο ρυθμό που να μην ξαναπέσει η χώρα σε μια κατάσταση δύσκολη. Θα έλεγα λοιπόν ότι ρεαλισμός και σύνεση είναι οι συστάσεις που πρέπει να κάνουμε. Πρέπει όμως και να σπρώξουμε, να πιέσουμε με κάθε μέσο για να ξεκινήσει η διαπραγματευτική διαδικασία. Και αυτό λαμβάνει η χώρα σε μια κατάσταση που ξέρουμε. Όπου η τρομοκρατία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Το ακούσαμε από όλες τι ερωτήσει και τη συζήτηση που έγινε. Δεν σας αρνούμε και το επαναλαμβάνω, διότι το είπα και στην αρχική μου παρέμβαση, ότι η θέση κατά της τρομοκρατίας είναι κοινή σε όλες τις χώρες του κόσμου. Σε αυτή την περίπτωση Μιλάμε για, μια, για διάχυτη τρομοκρατία με σύνορα ανοιχτά σε αυτή την περιοχή. Μεταξύ Μαλή και Αλγερίας είναι 1400 χιλιόμετρα τα σύνορα. Τε, τέτοιου είδους αποστάσεις έχουμε. Καταλαβαίνετε ότι η ανάπτυξη τρομοκρατία σε τέτοια περιοχή ε, είναι κάτι που μπορεί να μολύνει όλο τον κόσμο και πέρα από σύνορα και από συγκρούσεις και προβλήματα η Κίνα, η Ρωσία, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία έχουν την ίδια θέση. Απολύτω ίδια. Ακόμα και χώρε όπω η Αίγυπτος ε, που δεν ε, έχουν κρύψει την αντίδρασή του σε θετική δράση ο, ξέφρασαν όμως μεγάλη ανησυχία, μεγάλες ανησυχίες για την τρομο, ε, τρομοκρατία αυτή. Η τρομοκρατία από το Σαχέλ μήπως κατά κάποιο τρόπο μπορεί να επεκταθεί ε, και προς άλλες περιοχές. Υπάρχει μια επίγνωση που, την οποία πρέπει να εκμεταλλευτούμε για το καλό. Και το είδος των αποστολών που έκανα και κάνω έχουν αυτό το στόχο. Λέω, Εάν κάνουμε πονηριέ, θα μα ξεφύγει, αν δεν κινηθούμε σωστά και κάνουμε πονηριέ, θα ξεφύγει από τον έλεγχο η τρομοκρατία. Όταν λέω ότι είναι με τεράστιε. Τα όρια δεν είναι σαφή τη περιοχή. Μιλάω και για τι γειτονικέ περιοχέ, όπω είναι η Λιβύη. Ναι, υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Σα το λέω ξεκάθαρα. Εκφράζω την ανησυχία μου. Το στράτευμα το γαλλικό με την μεγάλη βοήθεια του Τσάντ προχώρησε, έκανε στατικές επιχειρήσεις που μπορούμε να θεωρήσουμε ως επιτυχής, όμως προφανώς σχεδόν όλα τα στατεύματα που ήταν αντίθετα εξαφανιστήκανε οι εχθροί. Σκορπιστήκαν, πήγαν στα βουνά, πήγαν στους γείτονες, πήγαν στη Λιβύη πιθανότατα τα εξωτερικά στρατεύματα, οι αντίπαλοι. Και αυτό είναι πρόβλημα το οποίο θα πρέπει απόλυτα εμεί να το αντιμετωπίσουμε. Να το αντιμετωπίσουμε πώ όμω. Και από άλλη σειρά ερωτήσεων που μου θέσατε, μπορώ να απαντήσω. Να αντιμετωπίσουμε με μια διαδικασία αναπτυξιακή που αντικαθιστά την οικονομία την παράνομη που ισχύει στην περιοχή. Το αναφέρατε με ευαισθησία, όμως πρέπει να θεμηθούμε ποια είναι η ποσοτική, ποσοτική σημασία του, των ναρκωτικών και του παράνομου εμπορίου, του λαθρεμπορίου, να προσθέσουμε και τις απαγωγές, εκβιασμούς, ε, ομήρους κλπ. Διότι τα τελευταίους μήνες ήταν ύψους ε, τα, λάφυρα για, ε, τα, λίτρα για, σε επίπεδο πολλών εκατοντάδων ε, χιλιάδων ευρώ. Λοιπόν αυτά τα προβλήματα δεν επιλύονται εάν δεν αντικαταστήσουμε την παράνομη υποστήριξη της ζωής των ανθρώπων με μια νομιμή οικονομία. Το πρόβλημα λοιπόν της μελλοντική ανάπτυξης είναι ένα πρόβλημα πρωταρχικής σημασίας, όπως σας υπενθύμησα και στην αρχική μου παρέμβαση. Είναι στο επίκεντρο των εργασιών μας. Δεν λέω σχεδόν όλη η δουλειά, το σημαντικότερο τμήμα της προσπάθειάς μας. αφορά αυτούς τους πυλώνες της ανάπτυξης που σας περιέγραψα. Έχουμε από τη μία πλευρά συντονισμό για παραγωγικές δομές, για τη δημιουργία μιας οικονομίας. Μην μη λησμονούμε ότι είναι ανεπαρκείς αυτές οι χώρες ακόμα και για βασικά πράγματα και για τα τρόφιμα. Ε, είναι αεροκατοικημένες ε, περιοχές, αλλά δεν έχουν αρκετά τρόφιμα, δεν έχουν επαρκή ενέργεια, δεν έχουν δομές welfare όπως τα αποκαλούσαμε, κράτους προνοίας, υγείας κλπ. για να μπορέσουν να κινηθούν. Πολλοί από εσά με ρώτησαν αν οι πολιτικές εξελίξεις και ο πόλεμος στη Λιβύη επιδίνωσαν την κατάσταση. Η απάντησή μου είναι ναι. Είναι προφανές. Υπάρχει μια ισορροπία, υπήρχε μια ισορροπία που διαταράχθη από αυτόν τον πόλεμο. Και γι' αυτό χρειάζεται δράση διεθνής για να αντιμετωπιστεί αυτό. Βέβαια, όλο αυτό, και εδώ αφορά μια άλλη σειρά ερωτήσεων, αυτό επηρεάζει λίγο το θέμα της ετερογένειας, της ποικιλομορφία εθνοτήτων, φυλών, κοινωνικών παραδόσεων. Εδώ εντάξει σημαντικό τμήμα είναι του ΑΡΕΓ. Δεν είναι ποσοτικά όμως το κυρίαρχο τμήμα. Μην το λησμονούμε. Είναι σαφές λοιπόν, όταν επιμένω στις διαπραγματεύσεις, σε αυτό προσπαθώ να ευνοήσω μια θέση ενοποιημένη, ενιαία από την πλευρά εκείνων που κατοικούν το Βορρά. Δεν είναι ένας στόχος κεκτημένος. Δεν είναι κάτι το κεκτημένο αυτό. Και αυτό πρέπει να γίνει, να επιτευχθεί με προσπάθεια. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας απαντήσω με αυτά που ρωτήσατε για το θέμα του Κατάρ, χρηματοδότηση κλπ. Υπάρχουν κάποια κουτσομπολιά, φήμες που ακούγονται, αλλά στοιχεία ε, ε, είναι πολύ περίπλοκο να συλλεχθούν για τη χρηματοδότηση από άλλες χώρες, για την τρομοκρατία. Είναι σαφές ότι αυτά τα ζητήματα Έχουμε ετοιμάσει απάντηση οργανική για τη μελλοντική ανάπτυξη. Πρέπει να μαζέψουμε χρήματα, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά από όλο τον κόσμο. Και εδώ τίθεται ένα πρόβλημα περίπλοκο. Υπάρχουν θέσεις, τοποθετήσεις διαφόρων χωρών, αρκετών χωρών, που θέλουν μια, να κάνουν μια παρέμβαση βοήθειας, αλλά με κάποιο τρόπο θέλουν και κάποιο είδος ιδιοκτησίας, ownership. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε μορφές ε, παρέμβασης που βγάζουν τα παλιά γραφειοκρατικά εμπόδια από τη μέση, αλλά μπορούν να δημιουργήσουν κάποιο ιδεώδη ανταγωνι... Ε, καλό ανταγωνισμό μεταξύ των τριών χωρών. Το μήνυμα που έδωσα στις διάφορες χώρες, τους Ρώσους, τους Αμερικανούς και τους Κινέζους είναι απλό. Είπα, έχετε συμφέρον. Να έχετε μια Αφρική που να μην έχει τρομοκρατία. Και για την ασφάλειά σας για τα τρόφιμα, για την ενεργειακή σας ασφάλεια, για την ασφάλειά σας όσον αφορά τις πρώτες ύλε στο μέλλον. Δεν έχετε συμφέρον να έχετε μια Αφρική που δεν είναι πλέον ένα στατόπεδο πεδίο της μάχης, αλλά ένα πεδίο συνεργασίας. Εκμεταλλευόμενος, όπως σας έλεγα, την κοινή τοποθέτηση κατά της τρομοκρατίας, θέλω να δημιουργήσω, να δημιουργήσουμε μια σύμπραξη ιδανικής ε, παρέμβασης, θετικής παρέμβασης. Χρησιμοποιηθεί η Αφρική σαν ένα πεδίο συνεργασίας και όχι σαν πεδίο μάχης. Βέβαια είναι πολύ ουτοπική αυτή η προσπάθεια θα έλεγα. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό ουτοπίας. Είναι ένα μήνυμα, πώς να το πω, ε, ευφυές, θα έλεγα αφελές ίσως, αλλά ξεκινά από μια βάση. Μπορεί να εφαρμοστεί όμως τελικά. Εκτός εντολής δεν μπορώ να δώσω απαντήσεις. Όπως για τις εντάσεις στην έρημο ε, και διάφορες αποστολές εκεί πρέπει να πω η εντολή που δόθηκε ε, κάποιες αποστολές δεν πέτυχαν να επιλύσουν τα προβλήματα. Αλλά αυτά τα ερωτήματα που εκτός της εντολής μου ε, και σωστό είναι να μην ξεπεράσω τα όρια της εντολής που μετέθη προσπαθώντας να απαντήσω σε αυτά που τα άλλα ερωτήματα που και δεν έχω καλύψει. Και τέλος φτάνω προς το τέλος διότι εξαντλείται, είναι περιορισμένος ο χρόνος μου. Ζητώ συγγνώμη που ομαδοποίησα τις απαντήσεις σε οικογένειες και δεν απάντησα μεμονωμένα σε κάθε προβουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση και υπάρχει μια κοινή ερώτηση που ετέθη, που ετέθη από πολλούς και αυτή αφορούσε την ευρωπαϊκή πολιτική έναντι της Αφρικής. Θέλω να πω ότι επιστρέφω στις εποχές που ήμουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τότε και στο μέλλον ίσως υπήρξαν, υπήρχε κάποια τοπική προσέγγιση. Να δημιουργηθεί αυτό ο δακτύλιο των φύλων. Όλες οι χώρες που είναι γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από Ευρώπη, από Λευκορωσία, Ουκρανία, μέχρι Μαρόκο, όλες οι χώρες να έχουν συμφωνίες, να έχουν σχέσεις και επαφέ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλα τα κεφάλαια, σε όλες κατηγορίες όλα, όλα εκτός από τους θεσμούς, everything but institutions, για να η, Ευρώπη να περιβάλλεται από αυτό που λέγαμε στη γνωστή η, ε, The Ring of Friends αποκαλούσαμε στη, δικό μας, στη δική μας ορολογία. Το δακτυλί, ο δακτύλιος των φίλων. Είναι οδυνηρό για μένα όταν ταξιδεύω σε αυτές τις χώρες και λέτε ότι είσαστε ο μεγαλύτερη χώρα, ο μεγαλύτερος επενδυτής, και είναι οι χώρε που μα ξέρουν καλύτερα και έχουμε ελάχιστε επαφέ μαζί του με αυτέ τι χώρε τι γειτονικέ. Αυτή, είναι η πραγματικότητα που είδα και αποκαρδίωσε. Αλλά πρέπει να το πω ότι ε, αυτό αισθάνομαι όταν συνομιλώ με κοσμό των χωρών. Ο κ. Σαλαφράγκα το έθεσε. Πρέπει να περάσει η βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση πέρα από τα όρια τη βοήθεια. Από τη φύση τη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να περιβάλλεται από δακτύλιο φύλων. Και αυτό κοστίζει πολύ λιγότερο από αυτό που κοστίζουν οι στρατιωτικέ παρεμβάσει. Που πρέπει να γίνονται καμιά φορά όταν ε, αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις στις οποίες οποίε μπορούσα να απαντήσω και αναλυτικά, όπως το ερώτημα που ετέθη. Αν η αλλαγή του κλίματος επηρέασε πολύ τις πτυχέ που ανέφερα, σίγουρα. Δεν είμαι ειδικό για το θέμα, αλλά όλοι μου λέγουν ότι τα ακραία φαινόμενα αυξήθηκαν, επιδεινώθηκαν. Μεγάλες περίοδοι ξηρασίας, λειψιδρίας, με πλημμύρες μετά, έχουμε μια επιδείνωση των ακραίων φαινομένων τα τελευταία χρόνια. Οπότε προφανώς και αυτό πιθανότατα επηρέασε την ε, κατάσταση στην περιοχή. Είδου, αυτά είναι τα ουσιαστικά σημεία και οι βασικές απαντήσεις που μπορώ να δώσω στις ερωτήσεις σας και σύντομα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να προσφέρει την εμπειρία της σε συμφωνία με τον ΟΗΕ, όπως αναφέρθηκε για την εκλογική διαδικασία να υπάρχει συνεργασία. Έχουμε μοναδική εμπειρία, πάρα πολλές χώρες, με πραγματική κληρονομιά και κατά την άποψή μου σε αυτή την περιοχή η διαδικασία που ξεκίνησε βοήθειας πρέπει να εντατικοποιηθεί σε αυτή τη φάση, διότι είναι μια ειδική περίπτωση αυτή τόσοι εκτοπιστέντες. Το πρόβλημα της κατάρτισης των εκλογικών καταλόγων είναι εξίσου σημαντικό με το πρόβλημα της ελευθερίας της προεκλογικής εκστρατείας και της μυστικής ψηφοφορίας στις εκλογές. Σε άλλες περιπτώσεις ήταν λιγότερο σημαντικά αυτά, αλλά σήμερα πρέπει να αναδιαργανωθεί μια ολόκληρη κοινωνία, η οποία κατακαιρματίστηκε. Πιστεύω ότι αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο που εκπροσωπείται εδώ από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων έχουν ένα ρόλο που ξεπερνά το υλικό πεδίο. Ε, έχουν ρόλο υποδειγματικό να παίξουν. Και η Αφρική χρειάζεται αυτό το όραμα. Και είναι κοντά μας, είναι η γειτονιά μας. Ε, έχουν ξεχάσει το παρελθόν δημιουργούνται, έχουμε συναισθήματα πως δημιουργούν αυτές οι χώρες που προσβλέπουν προς την Ευρώπη. Πρέπει να τη βλέπουν σαν φιλική, να τη βλέπουν θετικά. Να το βλέμμα από εδώ και μπρος, το βλέμμα μας να κοιτάει προς το μέλλον, όχι το παρελθόν και το βλέμμα εκείνων. Έτσι πρέπει να κινηθούμε, όχι μόνο στον οικονομικό τομέα, που χρειάζονται τα χρήματα, αλλά χρειάζεται και πολιτική κινητοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση. Πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Ευχαριστώ. Πρόεδρε Πρόντι, αγαπητέ Ρωμάνο, σε ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας. Συγγνώμη που έχω έρθει τόσο αργά. Είχα ένα πρόβλημα με την, ε, <laughs> με την έλευσή μου. Χρειάστηκα να βγω και από το αυτοκίνητο και να περπατήσω γιατί δεν προχώρησε τίποτα. Θα ήθελα όμως, Ρωμάνο Πρόντι, να σε ευχαριστήσω θερμά Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι όλα αυτά τα προβλήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού. Είναι απαραίτητο να καταλάβουμε ότι υπάρχει προϋπόθεση μεγαλύτερης ολοκλήρωσης, η προϋπόθεση του να αντιμετωπίσουμε τα κοινωνικά προβλήματα για να ξεπεραστεί το θέμα της τρομοκρατίας και του εμπορίου των ναρκωτικών και έχουμε ήδη την εμπειρία από προηγούμενες χώρες όπως το Αφγανιστάν και Παρ' όλα αυτά δεν καταλήξαμε στο αποτέλεσμα που θέλαμε. Το Αφγανιστάν τώρα παράγει 8 φορές περισσότερα ναρκωτικά από ό,τι στο παρελθόν. Γι' αυτό θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει καμία ασφάλεια, καμία, υπερπή, καμία υπέρβαση των προβλημάτων τρομοκρατίας και ναρκωτικών χωρίς τη διάσταση της ανάπτυξης. Και ελπίζω ότι αυτή θα είναι και η βάση επί της οποίας θα βασιστεί η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον για την ανάπτυξη και θέλω να σας ευχαριστήσω για το γεγονός ότι συζητήσατε μαζί μας και τονίσατε τον πιο ισχυρό ρόλο που πρέπει να αναλάβει η Αφρικανική Ένωση και ο στόχος ο δικός μας θα πρέπει να είναι να ευνοήσουμε αυτήν την συνεργασία των Αφρικανικών χωρών για την αντιμετώπιση των πραγμάτων αυτών πρέπει η στάση μας να είναι πραγματιστική χωρίς να απολέσουμε από τους οφθαλούς μας τους στόχους μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας είχαμε και πάλι μεταξύ μας. Πρέπει να πούμε ότι η εποχή του πρώτη ήταν στην Κομισιόν, ήταν η εποχή μιας τομής, μιας ε, ανανέωσης στην Κομισιόν. Ήταν ίσως η ωραιότερη εποχή που έχουμε γνωρίσει στην Κομισιόν και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και πάλι να είσαστε μαζί μας. Ευχαριστώ και τους καλεσμένους μας, οι οποίοι έχουν έρθει, τον κύριο Μπέλκα Σέμ, που τους συναδέλφους από την Αλγερία, το Μαρόκο και την Τινησία, που μας διευκρίνησαν και τις δικές τους θέσεις και μας τόνισαν ότι η σωστή κατεύθυνση είναι η κατεύθυνση η οποία θα πρέπει να βασίζεται στην κοινή δράση όλων μας. Ελπίζουμε λοιπόν θα μπορέσουμε όλα αυτά να τα κάνουμε πραγματικότητα. Θέλω να ευχαριστώ και τους διερμηνείς μας, οι οποίοι ξεπέρασαν τον χρόνο τους και τους ευχαριστώ που μας δώσαν την ε, ευκαιρία να περατώσουμε τη συζήτηση αυτή και σας εύχομαι καλό βράδυ σε όλους. Mm.